Uh, ladies gentlemen, I have the pleasure to this very interesting... Καλή σας μέρα. Προεδρεύω εγώ σήμερα και αντικοθιστώ την ε, πρόεδρο, την κυρία Ντινάλνη, η οποία θα παρακολουθήσει βέβαια τα γεγονότα. Ε, πρέπει να ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη όμως. Οπότε, καταρχήν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ. Εγκρίνεται. Ανακοινώσεις Πρόεδρου. Δεν υπάρχουν. Και έγκριση των πρακτικών τώρα των προηγούμενων συνεδριάσεων. Αν έχετε σχόλια, μέχρι αύριο το πρωί παρακαλώ. Αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα. Και τώρα, Περνάμε στη σημερινή μας συνεδρία. Είναι μια ακρόαση που έχουμε με εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς για την έξαρση της κρίσης του COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπως επίσης και πώς μπορεί να ανταποκριθεί η Ευρώπη με νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα. Προεδρεύω εγώ λοιπόν όπως σας είπα και αντικαθιστώ εδώ την πρόεδρο, την κυρία Τινάλη, η οποία θα παρακολουθήσει από ε, τηλεδιάσκεψη την ε, σημερινή συνάντηση και θα ήθελα, παρόλο που εγώ προεδρεύω, να δώσω το λόγο στην ε, Πρόεδρο να κάνει μια εισαγωγή. Οπότε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να προεδρεύσετε πρώτα απ' όλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπηρεσίε έκαναν ό,τι μπορούν για να διεξαχθεί ομαλά η συνεδρίαση αυτή και γι' αυτό υποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να του ευχαριστήσω όλου, του τεχνικού, του διερμηνεί και όλου. Η Προεδρία βέβαια με τους 7 ε, εμπειρογνώμονες και τα λοιπά είναι ήδη κάτι σπουδαίο που κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε κάποια τεχνικά θέματα, θέλω να τα αποφύγω όταν προεδρεύει κανείς δηλαδή εξ αποστάσεως, γι' αυτό σας ζήτησα να αναλάβετε την Προεδρία. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεδρίαση και σίγουρα θα διεξαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πρόκειται ε, για θέμα που αποφάσισαν οι συντονιστέ της Επιτροπής μας να ε, συζητήσουμε με την ακρόαση αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς, ποιε είναι οι συνέπειες ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία από την κρίση COVID-19 και τι με ποιο τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. που συμφωνούν ότι οι συνέπειες είναι τεράστιες, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάτι άλλο και σίγουρα το έχουμε ξανασυζητήσει και το συζητάμε είναι η επιβράθυνση αλλά και η ανάκαμψη που δεν θα ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες. Θα είναι διαφορετικά αυτά τα στοιχεία ανάλογα με τη διάρθρωση των οικονομιών, των χωρών και την επιμέρους απάντησή τους στην κρίση. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων για παράδειγμα, αλλά και άλλα. Όπως σας είπα και πριν, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, οπότε και οι απαντήσεις που έδωσαν διάφορες χώρες διαφέρουν μεταξύ τους. Θα πρέπει να μην τεθεί σε κίνδυνο όμως η νομισματική μας ε, πολιτική, να έχουμε τις σωστές απαντήσεις και οι απαντήσεις ε, αυτές να βοηθήσουν ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να επιδείξουμε ανθεκτικότητα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορες διευκολύνσεις που θα προχωρήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Οι εμπειρογνώμονες που θα λάβουν το λόγο σήμερα και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, σίγουρα θα μπορέσουν να μας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και στόχους που πρέπει να θέσουμε στο έργο μας, να μας ενημερώσουν και να μας αποφασίσουν τελικά να λάβουμε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές, ευχαριστώ και εσάς που προεδρεύετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Τώρα, πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω τους πρώτους τρεις ομιλητές, τον Πιέρ Ολιβιέ Γκουρινσάς, που είναι καθηγητής παγκόσμιας διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλι στην Καλιφόρνια. Δεύτερο, την κυρία Ντανιέλα Γκαμπόρ, η οποία είναι καθηγήτρια οικονομίας και μακροοικονομικών και τον Λέξ Χόχνταν, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν. Συμμετέχουν και τα μέλη βέβαια της Οικονομικής Επιτροπής στην ακρόαση αυτή και το κοινό βέβαια που παρακολουθεί online την συνεδρίαση αυτή. Στόχος του πρώτου αυτού πάνελ της ακρόασης είναι να συζητήσουμε την ανάλυση και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Επιπτώσεις στην οικονομία μας. Στα δύο πάνελ, μετά από μια μικρή εισαγωγή ε, του Πρόεδρου, θα υπάρξει ένας ε, γύρος παρεμβάσεων. Επτά λεπτά έχει στη διάθεσή του ο κάθε εμπειρογνώμονας. Θα ακολουθήσουν τρεις ερωτήσεις και απαντήσεις ανά γύρο. Δύο λεπτά για την κάθε ερώτηση παρακαλώ και να λέτε σε ποιον απευθύνεται η ερώτησή σας επίσης. Μετά από κάθε γύρο ερωτήσεων οι προσκεκλημένοι μας θα έχουν στη διάθεσή τους 8 με 10 λεπτά για να απαντήσουν στο πρώτο πάνελ και 10 με 12 λεπτά στο δεύτερο πάνελ, δεδομένου ότι έχουμε τέσσερις ομιλητές αντί για στο δεύτερο πάνελ. Επίσης, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που σας ε, δίνουμε. Να ξέρετε ότι θα έχουμε διερμηνία για τις πρώτες δύο ώρες. Μετά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση στα αγγλικά μόνο. Η διερμηνία υπάρχει στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα πολωνικά. Και εξυπηρετούν τη συνεδρίασή μας. Να ξέρετε ότι βασίζονται στην ποιότητα του ήχου και τη εικόνας όσων συμμετέχουν εξ αποστάσεως προκειμένου να σας βοηθήσουν να περάσει το μήνυμά σας όπως θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έχουν σταλεί για τη σύνδεση και για τον τρόπο που πρέπει να μιλάτε. Να ξέρετε ότι τηλεφωνικές παρεμβάσεις ή όταν δεν υπάρχει εικόνα δεν θα μεταφράζονται. Ζητούμε επίσης από τους ομιλητές να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα εφόσον αυτή καλύπτεται από τη διερμηνία. Σας συστήνουμε επίσης να μην διαβάζετε τις ομιλίες σας. Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε σημειώσεις και να βασίζετε σε αυτές και να μιλάτε ελεύθερα και σε κανονικό ρυθμό. Οι διερμηνείς σας ευχαριστούν πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας αυτή. Τώρα ξεκινάω λοιπόν με τον γύρο των ομιλητών και θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας για 7 λεπτά τον καθένα, όπως είπαμε. Και πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τον κύριο Πιέρ Ολιδιέ Γκουρισσάς, που είναι καθηγητής παγκόσμιας διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλε. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, πολύ χαίρομαι και είναι και τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσω τις αναμενόμενες επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, ξεκινώντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος ολόκληρος, χωρίς προηγούμενο μάλιστα, τουλάχιστον μετά από την μεγάλη ύφεση ξεκίνησε το Μάρτιο που μας πέρασε και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να ισοπεδώσουν την ε, καμπύλη της πανδημίας με διάφορα μέτρα που συνδύασαν με περιορισμούς που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις και με την επιβολή κοινωνικών αποστάσεων. Οι πολιτικές αυτές ε, βέβαια οδήγησαν σε κατάρρευση τόσο στη ζήτηση όσο και στην ε, προσφορά. Άρα λοιπόν καθοδική πορεία στην οικονομία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΣΑ, η δραστηριότητα σερικνώθηκε με 20 έως και 30% κατά τη διάρκεια των περιορισμών αυτών, δηλαδή της πάυσης της οικονομικής δραστηριότητας και η Ευρωζώνη αναμένεται να σερικνωθεί στο 9,1% φέτος. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ε, βέβαια οι αρχές είναι να δημιουργήσουν τα κατάλληλα δίκτυα ασφαλείας για να προστατεύσουν τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κάτι το οποίο απέτησε βέβαια μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις από τις δημοσιονομικές αρχές και συνδυασμό προγραμμάτων για την προστασία των εργαζόμενων, ε, αναβολή πληρωμής φόρων, ε, δάνεια με εγγύσεις προς τις επιχειρήσεις, ε, προσωρινά μέτρα και στοχευμένα βέβαια προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτές οι πολιτικές βέβαια μπορούν να είναι επιτυχές και έχουν όντως αποφύγει ευρύτερες απολύσεις. Οι πολιτικές αυτές όμως κοστίζουν κιόλα. Για την Ευρωζώνη ο ΩΣΑ, αναμένει ότι η σχέση του δημόσιου χρέους προς το ΕΠ θα φτάσει 104% από το 104% στο 121% το 2020, που είναι βέβαια για πρώτη φορά στην ιστορία τόσο χαμηλά τα επιτόκια και αυτό είναι που έχει βοηθήσει μέχρι τώρα την κατάσταση. Η κατάσταση αυτή όμως συγχρόνω πιέζει πάρα πολύ τις πιο ευάλωτες οικονομίες, αυξάνοντας τους κινδύνους για καθοδική πορεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανταποκρίθηκε έγκαιρα και αποφασιστικά στην απειλή αυτή ε, υιοθετώντα προσωρινά και στοχευμένα μέτρα όπω είναι το ΠΕΠ που πρόκειται για το πρόγραμμα αγορά στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημία για 1.350 δισεκατομμύρια, 11,3% δηλαδή του ΕΠ. Κάτι το οποίο ήταν πολύ βασικό και βοήθησε να σταθεροποιηθεί η αγορά και οι προσδοκίες. Τελικά βέβαια χρειάζεται μεγάλη δημοσιονομική αλληλεγγύη και οι τελευταίε ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα νέο μέσο ανάκαμψη, το Next Generation EU, με 750 δισεκατομμύρια ευρώ για ε, προσωρινά μέτρα ανάκαμψη, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει ακραίου κραδασμού που οφείλονται στην πανδημία. Τώρα βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις μπροστά μας. Και εδώ έχω να κάνω έξι παρατηρήσεις. Πρώτον, πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι ο λογισμός τους και η ρευστότητά τους επιδεινώθηκαν κατά πολύ κατά την πάυση της οικονομικής δραστηριότητα. Ε, πρόσφατα εγώ ανέφερα διάφορα στοιχεία έχοντας δείγμα από 17 χώρες, 14 από τις οποίες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκτίμηση είναι ότι 12% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαν να κινδυνέψουν μέχρι τα τέλη του 2020, ενώ συνήθως είναι 4,5% σε μια κανονική χρονιά. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι κυρίως εστίασης, ε, στέγασης, ε, πολιτισμού, ψυχαγωγίας, ε, λιανικό εμπόριο που είναι 5% της συνολικής απασχόλησης. Έτσι λοιπόν υπάρχει κίνδυνος και μην το ξεχνάμε αυτό να τοχεύσουν διάφορες επιχειρήσεις. Το κύμα αυτό λοιπόν ε, κινδύνου για τις επιχειρήσεις επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τράπεζες για παράδειγμα που είχαν κεφαλοποιηθεί πριν από την ε, κρίση αλλά βρίσκονταν ακόμα σε έφραυστη κατάσταση είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Με 3.000 δισεκατομμύρια δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη η αύξηση του κινδύνου αυτού για τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποσβεστεί με επιπλέον 250 δισεκατομμύρια. Αλλά αυτό ο κίνδυνο που υπάρχει είναι να αυξηθούν κατά πολύ τα μη ξεπηρετούμενα δάνεια, 2,1%. Ένα δεύτερο κύμα εξάλλου πολύ πιθανό να βρίσκεται ακόμα μπροστά μα. Έπειτα, υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία τη οικονομία αλλά και τη υγεία, που η αβεβαιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική ακόμα. Μέχρι τώρα ε, τα νοικοκυριά, για παράδειγμα, ε, αποταμίευσαν. Δεν ξέρουμε αν τώρα, όταν σταματάει δηλαδή ο περιορισμό, τα νοικοκυριά θα αρχίσουν να ξοδεύουν πολύ. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να είναι προσεκτικά και να μην ε, δαπανούν. Δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί λοιπόν η κατάσταση. Ίσως λοιπόν είναι πάρα πολύ νωρί να ξεκινήσουμε με δημοσιονομικά κίνητρα μεγάλης κλίμακος, να προστεύσουμε την απασχόληση και τις επιχειρήσεις όσο σιγά σιγά προχωράει η κατάσταση θα ήταν ίσως το πιο σωστό. Έπειτα, πολλοί λένε και πολύ σωστά ότι οι υπερβολικά γενναιόδορες πολιτικές ενισχύσεων θα μπορούσαν να εμποδίσουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε κόμμα κατά κάποιο τρόπο να γίνουν παραγωγικές. Εγώ θεωρώ ότι βράχει πρόθεσμα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι δεν θα έχουμε κάνει αρκετά, όχι ότι θα έχουμε κάνει υπερβολικά πολλά. Υπάρχουν ε, βέβαια το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, όπου υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Υπάρχει πάρα πολύ βεβαιότητα γενικότερα για το ποιοι τομεί θα θυχτούν πιο μόνιμα και ποιοι θα υποφεληθούν από τέτοια μέτρα. Είναι πολύ νωρί να αποφασίσουμε και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πέμπτον, συμφωνώ ότι δεν μπορούν ούτε θα έπρεπε να σωθούν όλες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την αναδιάρθρωση και τις διαδικασίες ε, ρευστότητας σε όλους τους κλάδους και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να περιμένουμε ότι οι επιπτώσεις από την πανδημία θα είναι ασύμετρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες εξαρτώνται πιο πολύ από τον τουρισμό για παράδειγμα και που κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από καθοδική πορεία της οικονομίας τους από ό,τι άλλες. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την οικονομική και την χρηματοπιστωτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζητούμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Ευρωζώνη που ίσως να χρειάζεται μάλιστα βοήθεια και από το μέσο Next Generation EU. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ντανιέλα Γκαμπόρ. Με ακούτε? Καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά συμμετέχω έστω και από μακριά στην ακρόαση αυτή. Αρχικά θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι η πανδημία COVID-19 φέρει αντιμέτωπα τα κράτη-μέλη με πάρα πολύ ε, βαθιέ αποπληθωριστικέ δυνάμει και ασύμετρου κραδασμού. Υπάρχουν ε, επομένω αυξήσει ε, στα νοσονομικά ελλείμματα. Το κόστο δανεισμού βέβαια παραμένει χαμηλό γιατί οι κεντρικέ τράπεζε είναι εγγυητέ και δημιουργούν αξιοπιστία. Θα ήθελα να απομυθοποιήσω τρία πράγματα. Ο πρώτο μύθο είναι ότι κεντρικέ τράπεζε ξεπέρασαν ε, το πεδίο της εντολής τους, ε, αναλαμβάνοντας τις ανάλογες ε, παρεμβάσεις στις αγορές των κρατικών ομολόγων θα αναφερθώ στην ΕΚΤΑ, αλλά αυτό αφορά και άλλα κρατημέλη. Υπονόμευσαν δηλαδή του μεσομικού κανόνε. Έχουμε τον ε, απόφαση του δικαστήριου τη Καλσρούη. Είναι ένα επιχείρημα ε, αντίστοιχο δηλαδή, που λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στα επίπεδα προκρίση. Ε, δηλαδή, η ΕΚΤΑ είναι αυτή η οποία θα έχει ω στόχο τη σταθερότητα των τιμών και τα κράτη-μέλη θα διεξάγουν δημοσιονομικέ και οικονομικέ πολιτικέ σύμφωνα με του ευρωπαϊκού κανόνε. Κατανομή δηλαδή των μακροοικονομικών εργασιών. Αν το δούμε μακρο οικονομικά είναι λάθος αυτό το επιχείρημα γιατί καθίσταται σαφές ε, αν δούμε την αλληλεπίδραση των ιδιωτικών ε, των ε, δομών και των οικονομικών πολιτικών ότι οι εξελίξεις στα οικονομικά έχουν ως αποτέλεσμα οι δημοσιομικές και οι νομισματικές πολιτικές να είναι κοινέ. Δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε πλέον. Αν λάβουμε υπόψη επίσης την μεγαλύτερη ε, αγορά, χρηματαγορά για ευρωπαϊκές τράπεζες και θεσμικού επενδυτές που είναι η αγορά των πράξεων επαναγορών, τρί, 7 7-3, δύο ε, είναι οι μεγαλύτερες χώρες Ευρωζώνης ε, που έχουν δανειστεί μέσω αυτών των πράξεων, Γερμανία και Ιταλία, με τη βοήθεια εγγύησεων. Και βέβαια έχουμε και τη δημιουργία ιδιωτική πίστη, που είναι το Σωμοτήρη των πράξεων των συναλλαγών τη ΣΕΚΤΑ που βασίζεται ε, στα κρατικά ομόλογα και στη μεσομονική πολιτική. Έχουμε υψηλότερε αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα κάνοντα ε, πιο ε, πανηρή την ιδιωτική πίστη. Η αγορά των ρέπο επίση και δημιουργία αλλά και μπορεί να καταστρέψει εύκολα τη ρευστότητα και κυβερνήσει, επηρεάζει τι συνθήκε δανειοδότη και τη μεσομονική πολιτική και στην Ευρωζώνη δημιουργεί μεγάλο προλέκτημα αυτό για τη Γερμανία και γι' αυτό και οι χώρε περιφέρεια. Ε, βλέπουν με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις και τα σπρέπτ ε, των γερμανικών ε, ομοσπονδιακών ομολόγων και δεν είδαμε να επεμβαίνει η ΕΚΤΑ. Το είπε και η πρόεδρος Λαγκάριστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ακρόαση ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η παρέμβαση. Χρειάζονται βελτιώσεις ε, σε αυτήν την ε, πολιτική. Οι ιδρυτές ε, δημιούργησαν μια δομή αλλά δεν είχαν λάβει υπόψη τους τις πολιτικές επιπτώσεις, ιδίως τις δομικές πιέσεις και τράπεζες να παρεύουν στις αγορές κρατικών ομολόγων. Επειδή αυξάνει η, ο λόγος δημόσιου χρέους ΑΕΠΑ και υπάρχει δυνατότητα, μάλλον η πιθανότητα νέας πίεσης ε, σε πιο ευάλωτα κρατικά ομόλογα, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Μέχρι στιγμή υπήρξε αυτοσχεδιασμό των κεντρικών πολιτικών με μη συμβατικά μέτρα πολιτική, ε, αλλά οι πόρου που ελέγχουν ε, έτσι έχουν ε, παγιώσει ένα δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο δημιουργεί αντιευρωπαϊκό αίσθημα. Στην Ευρωζώνη θα πρέπει η Νομισματική Ένωση να συνοδευτεί από τη Δημοσιονομική Ένωση, όχι μόνο για λόγου μεσονομική αλληλεγγύη, αλλά και γιατί η εναλλακτική θα ήταν μια τακτή έξοδο από το ευρώ, ιδίω αν οι φωνέ που ζητούν λιτότητα μετά την πανδημία γίνουν πιο δυνατές. Δεύτερος μύθος είναι ότι η Ευρώπη έχει θεσμούς που λειτουργούν καλά, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για να παράσχουν ένα δίκτυο ασφαλείας για τα κρατικά ομόλογα σε περίπτωση ή σε ε, κρίσεις ή σε καιρούς κρίσης. Υπάρχει και έκθεση αλμούνια για τα προγράμματα του Μηχανισμού Σταθερότητας και χρηματοπιστωτική ε, σταθερότητα στην Ελλάδα, που δείχνουν σημαντικέ αδυναμίε ε, στου θεσμικού μηχανισμού ε, για τη δημιουργία μηχανισμών προστασία ασφαλεία, backstop. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το κοινωνικό κόστο για του Έλληνε πολίτε. Δεν υπήρχαν στρατηγικοί στόχοι. Η προτεραιότητα δόθηκε συμφέροντα των μελών του Συμφουλίου Σταθερότητα και Μηχανισμού Σταθερότητα και όχι στην Ελλάδα. Και βέβαια υπήρξαν αυστηρά αντιπαραγωγικά μέτρα και όροι που επιβλήθηκαν ενώ ε, στις ιδιωτικές, ε, στον ιδιωτικό τομέα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Ακόμη και αν μπορούσαμε όμως να εφαρμόσουμε άμεσα τώρα τις συστάσεις Αλμούνια, ε, ένα μέρος μόνο του υψηλού δημοσίου χρέους θα μπορούσε να ελαφρυνθεί. Δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις κυκλικές πιέσεις ρευστότητας που δημιουργούν αυτές οι δομές που σας περιέγραψα, ιδίω εφόσον αυξάνεται και το βάρος του δημοσίου χρέους στην Ευρώπη και επίσης θα δημιουργηθεί και ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος ώστε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αντικυκλικές αντικυκλικού μάλλον με αντικυκλικό τρόπο του κραδασμού και να δώσει προτεραιότητα σε πράσινε δημόσιε επενδύσει και σε υποδομέ στο τομέα τη Γι' αυτό λοιπόν ε, το πρόγραμμα επιδοτήσεων τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματο EU Next Generation είναι ένα σημαντικό βήμα προ τη δημιουργία μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση. Αρκεί όμω αυτό. Και έρχομαι στον τρίτο μύθο που είναι ότι τα σχέδια ανάκαμψη από την πανδημία ε, είναι επαρκή. Μιλούμε για τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ινστιτούτο Μπρούγκελ περιμένει το 1 τέταρτο των επιδοτήσεων από το Next Generation EU να δαπανηθούν μέχρι το 2022. Από το 2020 έω το 2022 οι εθνικέ πολιτικέ είναι αυτό που θα πρέπει να υπομισθούν το βάρος της ανάκτησης, ότι της ανάκαψης. Θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να δώσει έμφαση στην οικολογική ανάκαμψη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν είναι θετικό που λέει ότι σκοπεύει το 25% των δαπανών να πάνε σε φιλοπεριβαλλοντικές δαπάνες. Οι προπάθειες θα πρέπει όμως να διευρυνθούν ε, για την πρόθεση βιώσιμων ε, ε, οικονομικών και την υποστήριξη των πράσινων κεντρικών τραπεζών. Παραδείγματο χάρη, η ΕΚΤ ε, στηρίζει του φορεί τη αγορά χωρί όμω ε, να συνδέει αυτό με όρου περιβαλλοντικού, φορολογικού ή εξόφληση. Ε, στη συνεχή δηλαδή να επιδοτεί δράσει με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα και έτσι δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ε, ποιοι θα ήταν οι στόχοι. Θα να ε, να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αρχίσει να θέλει να αγαπά τον καφετή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πληθωρισμό. Έχουμε τον ορισμένο δίκτυο τιμών καταναλωτού που αγνοεί το ε, αποτύπωμα άθρακα των αγαθών και των υπηρεσιών. Ε, επίσης θα πρέπει να είναι πιο πράσινες οι πολιτικές, ε, της ε, νομισματικές πολιτικές και ενέργειες της ΕΚΤΑ, να μην υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση στα πράσινα περισσιακά στοιχεία. Θα πρέπει να προωθούνται τα πράσινα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να μην έχουμε απλά ένα προσωπείο, ένα ψευδοπράσινο προσωπείο και πολιτικές τέτοιες, αλλά να αντιμετωπιστούν βιώσιμα τα προβλήματα. Και επίσης θα πρέπει να αποφασιστεί και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο ποιε είναι οι γενικέ πολιτικέ, οι οικονομικέ πολιτικέ που θα πρέπει να στηρίζει η ΕΚΤΕ. Στο άρθρο 11 τη ε, Συνθήκη για τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η περιβαλλοντική προστασία ξεκάθαρα σε σχέση και με το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων τη Κεντρική ε, Τράπεζα, που είναι ευρύτερο από την νομισματική πολιτική. Θα αποτελούσε την πολιτική νομιμοποίηση για τη δημιουργία ενό μηχανισμού ασφαλεία ανεφόρων ε, για τι πράσινε αυτέ επενδύσει και αυτό θα δημιουργήσει σημαντικό κέρδο σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κυριαρχία. Και για να ολοκληρώσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταθεροποιεί με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να επιταχύνει ω το δυνατόν περισσότερο το έργο τη ό,τι αφορά στρατηγική για, μια ανανεωμένη, για ανανεωμένα βιώσιμα οικονομικά. Πρέπει να έχουμε καλά καθορισμένη ταξινομία για πράσινε και καφετιέ δραστηριότητε και μέτρα προληπτική εποπτεία ε, που θα καθοδηγούνται ακριβώ από την ταξινομία ώστε η ιδιωτική χρηματοδότηση των καφετιών δραστηριοτήτων να μην υπονομεύσει τι πράσινε επενδύσει. Επόμενο ομιλητή. Έχετε 7 λεπτά. Η κυρία Alex Χόχτεν. Mr. Hochstein, could you please press the speak button? Thank you. Can I be here? Με ακούτε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω στην ακρόαση αυτή. Η πανδημία COVID-19 ήταν καταρχάς ένα πρόβλημα υγειονομικό. Ωστόσο, όταν ε, φάνηκε ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί απόλυτα ο ιός, ε, χτύπησαν την πόρτα και οι οικονομικές επιπτώσεις. Προκειμένου λοιπόν να μειώσουμε την πίεση που δεχτήκαν οι υγειονομικοί ε, υγειονομικό πορέα, ο υγειονομικό κλάδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάστηκε να επιβληθούν διάφορε μορφέ εγκλισμού. Και αυτό προκάλεσε μια ασυμμετρική, ένα ασυμμετρικό κλειδονισμό στην ε, αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, ενιαία αγορά. Και ε, παράλληλα είχαμε και ασυμμετρικού κλειδονισμούς στον εφοδιασμό εντό των χωρών. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μάλλον ευρεία συνένεση σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική που χρειάζεται για να τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία, λαμβάνοντα υπόψη την έλλειψη προφανώ εμβολίου και φαρμάκων. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει να κάνει με την παροχή υποστήριξη στο εισόδημα και στην ε, ρευστότητα και στην ε, γεφύρωση χρηματοδοτήσεων για νοικοκυριά και εταιρείε με ε, Κυβερνητικέ εγγύησει, ε, κρατικέ εγγύησει, Για να επιτρεχθούν λοιπόν αυτές οι πολιτικές σε ό,τι αφορά του κανόνε τους κανόνες για την χρέωση που έχουν οι χώρες. Ε, κάποιες ευρωπαϊκές λοιπόν, κάποιες ευρωπαϊκές, κάποιοι ευρωπαϊκοί κανόνες και τραπεζικές εφαλαιοκές ε, προδιαγραφές χαλάρωσαν. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν θα αποτρέψει απόλυτα μια βαθιά ύφεση. Βρισκόμαστε στη φάση που σιγά σιγά οι χώρες προσεκτικά βγαίνουν από το lockdown. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτό συμβαίνει μια στιγμή που ο ιός δεν έχει ακόμα ε, καταπνιχτεί. Ε, ένα σενάριο που θα εμπεριέχει διάφορα lockdown στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί. Γι' αυτό λοιπόν οι οικονομίες δεν έχουν μπει αυτό που θα αποκαλούσαμε τη φάση ανάκαμψης και θεωρώ ότι αυτή η φάση μπορεί να ξεκινήσει μόνο τη στιγμή που μπορούμε με σχετική βεβαιότητα να αποκλείσουμε ενδεχόμενο μελλοντικού lockdown. Όταν ο κορονοϊός, για παράδειγμα, θα θεωρηθεί ότι είναι υποέλεγχο. Η εφαρμογή λοιπόν τέτοιων πολιτικών ανάκαμψης στην παρούσα φάση έχει τον κίνδυνο να είναι μη αποτελεσματικέ γιατί θα είναι πρώιμε. Στην παρούσα φάση μπαίνουμε στην επόμενη φάση ελαγχού του ιού. Εξακολουθούμε να δερχόμαστε φάση κρίσης. Η αποτροπή νέων lockdown θα πρέπει να αποτελέσει τον πρώτο στόχο όλων των πολιτικών στην παρούσα χρονική στιγμή. Αυτό μόνο σε συνδυασμό Προφανώς με το άνοιγμα της οικονομίας και την ε, εκ νέου λειτουργία της έννοιας αγοράς. Αν οι χώρες θέλουν να περιορίσουν τον ιό με συντονισμένες δράσεις, με τέτοιες πολιτικές ε, ελέγχου ανείχνευσης και καραντίνας. Στην παρούσα φάση, τα νοικοκυριά, οι εταιρείε, οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις όλος ιδιαίτερος χρησιμοποιούν ε, προσωρινέ λύσει και δανεισμό. Και καλά κάνουν. Οι κυβερνήσει πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελέγξουν τον ιό, να περιορίσουν την ε, οικονομική ύφεση. Αλλά εδώ θα βάλουμε τελεία και θα πούμε όχι παραπάνω, τίποτα παραπάνω. Η δημοσιονομική πειθαρχία για το σκέλος που δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό θα πρέπει να διατηρηθεί σε ό,τι αφορά τους προπολογισμού. Γιατί να θυμηθούμε ότι ήδη πριν το ξεσπασμά του κορονοϊού, σε κάποιες περιπτώσεις ε, τα επίπεδα κυβερνητικής ε, χρέωσης ήταν προβληματικά. Και το ξέσπασμα του κορονοϊού προφανώς επιδίνωσε την κατάσταση και έφερε πιο πολλές χώρες στον κατάλογο των χωρών με προβληματικό κρατικό επίπεδο χρέωσης και αυτό προφανώς θα συνεχιστεί ω τάση. Η συνέπεια λοιπόν είναι ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση, σε μια λεπτή θέση. Η χρέωση, η κυβερνητική χρέωση, η κρατική χρέωση σε κάποιες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρώ μπορούν να διατηρηθούν μόνο με πολύ χαμηλά επιτόκια, όπως έχουμε στην παρούσα φάση. Και η έκτη λοιπόν αναγκάζεται να δράσει ως ε, παράγοντας ε, για την καμπύλη απόδοση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και έτσι ουσιαστικά βρίσκεται παγιδευμένη σε μια πολιτική με επικέντρωση στο χρέος. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτελέσει την εντολή τη και ενδεχομένω ε, μακροπρόθεσμα να έχει σοβαρέ επιπτώσει σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, την χρηματοοικονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ίδιου του ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν η προτεραιότητα της πολιτικής ε, στην έναρξη αυτή της φάσης ανάκαμψης, όχι ακόμα, όταν θα ξεκινήσει η φάση ανάκαμψης, θα πρέπει να είναι να α, μπορέσουμε να ξαναγεμίσουμε τα αποθέματα και να περιορίσουμε το επίπεδο δανεισμού και χρέωση από τα νοικοκυριά, τις τράπεζες, ε, τις εταιρείες και τις ε, κυβερνήσεις, Οι πολιτικέ οι οποίες ε, στην φάση αυτή θα επικεντρωθούν βασικά στην ε, παροχή κινήτρων σε ό,τι αφορά την ε, ζήτηση και την ανάπτυξη, θα έχουν προσμένα αποτελέσματα αν δεν υπάρχει πρώτα αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και επιπλέον δεν θα μειώσουν καθόλου τις ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και την κρατική χρέωση για το ευρώ και για την έκτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το... να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Δύο λεπτά παρακαλώ η καθερώτηση. Και να λέτε ξεκάθαρα σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας παρακαλώ. Μην ξεχνάτε επίσης να πατάτε το κουμπί ομιλία, speak, για να μπορέσετε να μιλήσετε. Ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο λοιπόν. Δύο λεπτά είπαμε ο καθένας για ερώτηση. Ο κύριος Γιώργος Κίρτσος παρακαλώ εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι από την Ελλάδα και άκουσα τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, θέλω να ρωτήσω για το δημόσιο χρέος. Είναι σαφές ότι το επίπεδο χρέους αυξάνεται. Στην Ελλάδα, από το 175% του ΕΠ, πηγαίνει στο 195, ίσως και στο 200% του ΕΠ. Οπότε η ερώτησή μου είναι, σύμφωνοι. Και η Ιταλία βρίσκεται σε αντίστοιχο πρόβλημα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, την επομένη της κρίσης, τι θα γίνει με τη βιωσιμότητα του χρέους. Γιατί αφενός μεν αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις πολιτικές που χρησιμοποίησαμε κατά το παρελθόν γιατί κοινωνικά και πολιτικά είναι απαράδεκτες. Η ερώτησή μου απευθύνεται και στους τρεις εμπειρογνώμονες, παρακαλώ. Είπατε και στους τρεις ομιλητές, απευθύνεται η ερώτησή σας. Έτσι είπατε κύριε Κίρτσο. Ναι, καλώς. Δεύτερη ερώτηση. Εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Σούστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που περιγράψαμε πολύ σωστά είναι το εξής, ότι σε μια τέτοια ε, βρισκόμαστε σε μια ε, πολύ περίεργη και εκθετή οικονομική κρίση, η οποία θα εμαθενθεί και Υπάρχουν κλειδονισμοί και στην πλευρά της προσφοράς και τη ζήτηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ασυνηθιστό. Και το βάθο ε, τη κρίση είναι πρωτόγνωρο. Πώ θα βγούμε λοιπόν από την κρίση αυτή. Σωστά τονίσαμε ότι βρισκόμαστε σε φάση που προσπαθούμε ακόμα να περιορίσουμε τη ζημιά. Το πρόβλημα όμως και το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς θα δώσουμε κίνητρα εκ νέου στην ε, οικονομία. Μία ερώτηση λοιπόν να κάνω προς τον κύριο Γκούριντσα. Είπατε στην ομιλία σας ότι είναι δύσκολο ότι δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε υπερβολικά όλες τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Δεν θα είναι δυνατό αυτό. Τι γίνεται με το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θέλω, θέλει να ε, εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το δεύτερο ήμιση του έτους ποιοι είναι τα κριτήρια για να επενδύσουμε στα σωστά πράγματα και κατά δεύτερον, τι γίνεται με τους τομείς εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν καν να υποστηριχθούν όσο ακόμα είναι παρόν ο ιός, όπως ο τουρισμός για παράδειγμα, όσο δεν επιτρέπεται για παράδειγμα να γίνονται σωστά ταξίδια, πώς θα προωθηθούν αυτοί οι τομείς. Πώς θα πάει κανείς στα εστιατόρια κτλ. Είναι όλα αυτά πολύ δύσκολα Πόσο διαφοροποιημένο λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα οικονομική ενίσχυση. Μία δεύτερη ερώτηση προ την κυρία Ντανιέλα Γκάμπορ. Είπατε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να ασκήσει πολιτική οικολογική. Αυτό συγκεκριμένα τι σημαίνει. Γιατί στην παρούσα φάση η ΕΚΤ πλημμυρίζει τις αγορές με χρήμα για να διατηρηθεί στο βαθμό του δυνατού η ρευστότητα. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει τέτοια διαφοροποίηση στην πολιτική αυτή. Και προς τον κύριο Χόχταϊν. Να κάνω την εξή ερώτηση. Ποια είναι αυτά τα τμήματα του προπολογισμού που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό, στα οποία μα είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία. Και πώς μπορούμε να φροντίσουμε, γιατί δεν μας είπατε πότε ακριβώς θα είναι η χρονική στιγμή αυτή, από πότε θεωρείτε ότι ξεκινάει η φάση της ανάκαμψης και μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που κάναμε το 2010 να βάλουμε δηλαδή υπό επιπλέον πίεση την οικονομική κατάσταση στις ε, χώρες. Ευχαριστώ και δύο ερωτήσεις λοιπόν έχουμε για κάθε ομιλητή και θα ήθελα να συνεχίσουμε με τον ε, κατάλογο των ομιλητών μας. Το λόγο έχει ο καθηγητής Γκουρανσά. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα μέρο της πρώτης ερώτηση και σε ένα μέρο της δεύτερης για τη βιωσιμότητα του χρέους. Οι εκτιμήσεις που έχουμε όλες για τα επιτόκια που θα παραμείνουν χαμηλά για διαρθρωτικούς λόγους για αρκετό καιρό ακόμα. Οπότε αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με το δημογραφικό ζήτημα, με την χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας, με τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία κλπ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα αυξηθούν τα πραγματικά επιτόκια σύντομα. Κάτι το οποίο μας δίνει περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε την βιωσιμότητα του χρέους με σοφό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αλλάζουμε τη συζήτηση και αρχίζουμε να συζητάμε πότε θα αυξήσουμε ε, τους φόρους για παράδειγμα. Το λάθος που έγινε το 2010 με την κρίση του δημοσίου χρέους ήταν ε, ακριβώς ε, αυτή, λάθος. Όσον αφορά τώρα με την, για την ανακατανομή και πώς θα ξεχωρίσουμε τις επιχειρήσεις που είναι φερέγγες από εκείνες που κινδυνεύουν κτλ. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ στις παρατηρήσεις μου, ότι αυτό είναι ο κίνδυνος. Στο στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό τόσο πολύ. Πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι προς τις επιχειρήσεις, ακόμα και αν στο μέλλον ε, χρειαστεί να ζητήσουμε πίσω κάτι από τα κέρδη για παράδειγμα. Οι επιχειρήσεις που θα ε, πάρουν στήριξη, κάποιες θα μπορέσουν να επιστρέψουν κάτι, κάποιες άλλες όχι. Πάντως, δεν πρέπει να κόψουμε τη στήριξη πολύ νωρίς. Κάποιοι κλάδοι, ακούσαμε για τον τουρισμό και υπάρχουν και άλλοι βέβαια, ε, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο για να είμαστε σε θέση να τους επαναφέρουμε σε βιώσιμη κατάσταση, ό,τι και αν κάνει το κράτος. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας επίσης. Ευχαριστούμε κυρία Γκαμπόρ. Ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Έθεσε ένα πολύ σημαντικό θέμα ο, ο μιλητής για τους ακαδημαϊκούς, δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε την βιωσιμότητα του χρέους. Και η ειλικρινή απάντηση είναι ότι πια δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε τα μέσα για να κατανοήσουμε ικανοποιητικά τι είναι βιώσιμο, κυρίως μετά τους κραδασμούς αυτούς της πανδημίας. Ε, ξέραμε πριν, βάζαμε κάποια αναλογία, ε, χρέους τώρα πια δεν ισχύει καλά-καλά. Οπότε Πρέπει να αλλάξουν τα κριτήριά μας για τη βιωσιμότητα και να δεχτούμε ότι ζούμε σε μια νέα κατάσταση ε, εξαιτία της πανδημίας. Θα μας πάρει χρόνο τα ελλείμματα στους προπολογισμούς παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ιδιαίτερα υψηλά και το χρέος επίσης. Οπότε η απάντηση στο τι πρέπει να κάνουμε, όπως είπε και ο κύριος Γκουρίνσας πριν από λίγο, είναι ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη δημοσιονομική ε, πειθαρχία, τη λιτότητα, δημοσιονομικά μέτρα κτλ. Όχι. Ανάπτυξη πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, να φροντίσουμε για τις δημόσιες επενδύσεις, την πράσινη ανάκαμψη που μπορεί να βοηθήσει στην ε, απασχόληση. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε τις κεντρικές τράπεζες και οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να κάνουν αυτό που είπε και ο καθηγητής Χόκτουιν, δηλαδή στοχευμένα μέτρα ώστε τα επιτόκια για το δημόσιο χρέος να παραμείνουν χαμηλά και ε, το δημόσιο χρέος και η αποπληρωμή του επίσης. Διαφωνώ με τον καθηγητή Χόκτουιν όσον αφορά την μείωση του χρέους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, γιατί αυτό θα αυξήσει την επιβράδυση της οικονομίας αντί για το αντίθετο. Όσον αφορά τώρα το πρασίνισμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η πρόεδρος Λακάρτ ήδη είπε ότι στην επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΚΤ θα συζητήσουν για τις εξασφαλίσεις, τι θα δέχονται σαν εξασφαλίσεις, ε, μη συμβατικά μέτρα πολιτικής και κατά πόσο θα ε, δώσουν ευνοϊκή μεταχείριση ή όχι σε πράσινα ή μη πράσινα ομόλογα. Η ταξινόμηση λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει γρήγορα γιατί αυτή θα μας βοηθήσει να καταχωρήσουμε τις επενδύσεις σε πράσινες ή μη είναι πολύ σημαντικό το πρασίνισμα των επενδύσεων. Θα πρέπει να είναι πιο ακριβώς ο διανισμός εφόσον υπάρχουν εξασφαλίσεις που βασίζονται σε μη ε, πράσινα στοιχεία. Το ίδιο και για τα εταιρικά ομόλογα που έρχονται από κλάδους υψηλής έντασης άθρακα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χοκτών τώρα για να απαντήσει στις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, για την πρώτη ερώτηση όσον αφορά το χρέος και πώς να μειώσουμε τα επίπεδα χρέους. Για αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να τονίζουμε πολύ και καθόλου τη βιωσιμότητα του χρέους, η πεποίθησή μου είναι ότι τα χαμηλά επιτόκια βοηθούν στην βιωσιμότητα του χρέους. Δηλαδή εκεί οφείλεται η βιωσιμότητα. Νομίζω όμως ότι τα σημερινά επίπεδα, τα χαμηλά επιτοκίου, τα πιο χαμηλά εδώ και 35 χρόνια, δεν θα μπορούν να βοηθήσουν για πολύ ακόμα. Και θα έλεγα μάλιστα ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αν αποδεχτούν λάθος τα μέτρα, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Πώς θα περιορίσετε το χρέος σε πιο βιώσιμα επίπεδα μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν, θα έλεγα, πέντε τρόποι για να το πετύχει κανείς αυτό. Ένα είναι να διατηρηθούν χαμηλά τα επιτόκια. Είναι οι τρέχουσε πολιτικές της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ελέγχει τα επίπεδα χρέους. Εξήγησα ότι πρέπει να βασιζόμαστε λιγότερο σε αυτό, κατά τη γνώμη μου. Μετά έχουμε την ανάπτυξη. Για να βγει κανείς από το αλλά δεν πρόκειται για μέσο πολιτική, πρόκειται για το αποτέλεσμα κάποιων μέτρων πολιτικής. Όσον αφορά το New Generation EU και την πράσινη ανάκαμψη, θα έλεγα ότι αν προσπαθείτε να ακολουθείτε μια πολιτική για την μέγιστη δυνατό ανάκαμψη, τελικά αν αντικαταστήσετε δηλαδή την ικανότητα των ορυκτών για ανάπτυξη από την πράσινη ικανότητα, δεν βοηθάτε να ε, μειώσετε το χρέος σας ε, μακροπρόθεσμα, γιατί δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη έτσι. Διακόπτει ο πρόεδρος, ο κύριος Έπινγκ. Δεν έχουμε χρόνο, οπότε παρακαλώ σύντομα. Συνεχίζω κύριε Σχοφτάουν. Οι άλλες πολιτικές είναι η λιτότητα και η αναδιάρθρωση. Πράγματα τα οποία φυσικά θα πρέπει να συμφωνηθούν μέσα σε ένα νέο πλαίσιο. Για τη δεύτερη ερώτηση τώρα, σύντομα. Ποια είναι, ποιο είναι το κομμάτι εκείνο που δεν έχει να κάνει με την πανδημία. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα και του Πρόεδρου Συνέδρου του κ. Έπιν και του μιλητή. και... Διακόπτη ο κύριος Χοχτάν. Ο κύριος Γκαρικάνο. Δύο λεπτά παρακαλώ είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έπινγκ. Καταρχάς, στον πρώτο μιλητή, τον κύριο Γκουρίνσα για τη συνολική ζήτηση και για τις δαπάνες από τα νοικοκυριά. Τι θα γίνει αν έχουμε υπερβολικέ δαπάνε από τα νοικοκυριά, ε, κεντρικέ τράπεζε, ε, υπάρχουν τα σωστά κίνητρα. Επειδή και το χρηματοψηφιακό σύστημα εξαρτάται από την ευθυνή πίστη. Το δεύτερο για το σχέδιο ανάκαμψη ε, ανθεκτικότητα. Λέτε ότι δεν είναι πολύ φιλόδοξο, έρχεται αργά. Ε, και ποια είναι η δική σας άποψη και σε σχέση με το σχεδιασμό του και την αναλογία επιδοτήσεων και δανείων. Και τι αποδείξεις έχουμε δει. Πρώτη προτεραιότητα στο χρέος και μετά στην ανάκαμψη. Πώς το εξηγείτε. Είδαμε πώς πάλεψε να πετύχει τον Ιωτήλο Ρούζβελτ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω έχουμε το αντίθετο σχήμα. Γιατί δεν θα έχουμε καθόλου ανάπτυξη αν προσπαθήσουμε πρώτα να αποπληρωθεί όλο το χρέος. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης, κύριε Γκούρινς. Ευχαριστώ τον κύριο Γκαρικάνο, λέει ο πρόεδρος. ID. Γκούναρ Πεκ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι τον κύριο Γκουρανσά. Θα ήθελα επίσης και ο κύριος Χουχτάιν να απαντήσει. Κύριε Γκουρανσά, είπατε ότι ίσως υπάρξει κίνδυνος να δοθούν υπερβολικά πολλά οικονομικά κίνητρα πολύ νωρίς. Και υπάρχει κίνδυνος με τις τομεκές πολιτικές. Να μην δώσουν εκεί που πρέπει το βάρος. Θα ήθελα να μας πείτε οι κίνδυνοι που βλέπετε να σχετίζονται με αυτό που έγκυται. Και επίσης ο κύριος Χοφτάιν για αυτά τα δύο. Τι έχει να μας πει, γιατί νομίζω ότι σχετίζονται με τις δικές του προειδοποίησεις ε, ως προς την έκτα, ότι ίσως προχώρησε πολύ στο μονοπάτι της ποσοτικής χαλάρωσης ε, για να αντιμετωπίσει την άνοδο του πληθωρισμού με συγκεκριμένα μέτρα. Και έχω και μια ερώτηση προς την κυρία Γκαμπόρ, που φαίνεται να μας είπε ότι δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη κάποια πράγματα στις συνθήκες ούτε και στην εντολή τη ΕΚΤ περιλαμβάνονται και υπάρχουν κίνδυνοι ή θα υπήρχαν κίνδυνοι άτακτης έξοδου κάποιων κρατών μελών, την Ευρωζώνη κατάρρευσε ενδεχομένω και του ευρώ. Και καταλήξατε στο ότι η συνθήκη πρέπει να διορθωθεί προς αυτό. Αν η πρόθεση είναι να έχουμε αυτή την τροποποίηση της συνθήκης για να είναι όλα νόμιμα πέραν πάσης αμφιβολίας, θα συμφωνείτε τότε ότι αυτή η νομιμότητα των μέτρων να τίθεται από αμφισβήτηση στην παρούσα χρονική στιγμή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά έξι ερωτήσεις είχαμε για δύο από τους τρεις ομιλητές. Θα παρακαλέσω τους ομιλητές να δώσουν σύντομες απαντήσεις, διότι σε κάθε γύρο έχουμε περισσότερες από τις προβλεπόμενες ερωτήσεις τελικά. Ο κύριος Σάιν, ο πρώτος, εν συνεχεία ο κύριος Φαχντά και η κυρία Γκαμπορ, εν κατακλείδη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. γιατί νομίζω οι ερωτήσει Γκαριγκάνο και Μπέκ σε έναν βαθμό αλληλεπικαλύπτονται. Το ερώτημα είναι αν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι περιορισμοί ε, τη προσφορά είναι ε, μεγαλύτεροι από τη συζήτηση το ανάποδο. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μείωση στην ζήτηση και αυτό ήταν ο βασικό παράγοντα μέχρι τώρα. Αυτό που δεν το γνωρίζουμε ακόμα είναι πόσο θα ανακάμψει και πόσο γρήγορα θα ανακάμψει η ζήτηση. Και γιατί λέω ότι είναι ο παράγοντα ο βασικό που περιόρισε τα πράγματα, είναι ότι υπήρξαν πιέσει, οι οποίε όμω μειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ίσως κάποιοι ε, αρχίσουν να θελήσουν να ξαναξοδεύουν γιατί πολλά νοικοκυριά αποταμίευσαν πολλά ποσά ε, αυτή την περίοδο. Ε, ε, Βγαίνοντα λοιπόν από την απομόνωση και από την καραντίνα, έχουμε το ερωτηματικό τι θα κάνουν τα νοικοκυριά. Αποφασίζουν να, να δαπανίσουν πολλά ποσά σε αγαθά διαρκεία ή άλλα αγαθά τα οποία δεν είχαν μπορέσει να αγοράσουν του τελευταίου δύο-τρει μήνε. Αν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε μεγάλη ανάκαμψη της ε, ζήτηση. και τότε ερχόμαστε στην προσφορά. Οι επιχειρήσει πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά στο περιβάλλον. Και όπω είπε και κάποιο ομιλητή πριν, Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Αν φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την ε, φάση, εγώ περιμένω οι νομισματικές αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει και ανήκει στο πεδίο της εντολής τους, δηλαδή να προσπαθήσουν να περιορίσουν ε, πιέσει στη τιμές αν είναι πολύ μεγάλες και αν ε, υπερβαίνεται συστηματικά εντολή τους. Αλλά ίσως αντί να χρησιμοποιηθεί δημοσιονομικό κίνητρο, όχι νομισματικό, να γίνει μια προσπάθεια να γυρίσουμε στο τέταρτο εξάμεινο του 19 για παράδειγμα ε, την οικονομία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει και το έργο των μοσαμικών αρχών και των νοσηματικών αρχών θα είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί θέλουν τώρα να διατηρήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά ταυτόχρονα να τηρήσουν και την εντολή που έχουν ό,τι αφορά τις τιμές και εκεί θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ευχαριστώ. Κύριος για δύο ερωτήσεις τώρα. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ πολύ για την τελευταία ερώτηση. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε ο καθηγητής Γκουρανσά. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, τις, ε, με τη ζήτηση και αν δεν λειτουργήσουν τα κίνητρα και είναι αντιπαραγωγικά. Η δική μας ε, η εμπειρία από διακριτική παροχή κίνητρων τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι θαρρυντική. Αυτό για το πρώτο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά το χρέος, μετά το τέλος της πρώτης φάσης της κρίσης, όταν είναι πλέον υπό έλεγχο κορονοϊός και δεν φοβόμαστε πλέον κατάρρευση των συστημάτων υγείας, τότε, σε αυτή τη χρονική στιγμή, έχουμε αυξημένο χρέος. Και χρησιμοποιούμε αυτά τα αποθέματα ασφαλείας, τα λεγόμενα buffer. Και υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθούν αυτά τα buffer, αυτά τα αποθέματα ασφαλείας, να έχουμε πολύ υψηλό χρέο και αρχίσουμε ταυτόχρονα να τονώνουμε, να προσπαθούμε να τονώσουμε την οικονομία ο κίνδυνος που δημιουργείται είναι να μην λειτουργήσουν αυτά τα κίνητρα. Γιατί δεν μπορούν να επενδύσουν λόγω του ψηλού χρέους που έχουν οι επιχειρήσει στα νοικοκυριά. Και έτσι δεν θα λειτουργήσει. Να απαντήσω κάτι που δεν μπορούσα να απαντήσω στον πρώτο γύρο ερώτα απαντήσεων τι σχετίζεται και τι δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό. Σχετίζεται φυσικά με τον κορονοϊό ιατρική δαπάνη και οι σχετικές δαπάνες για την εισοδηματική στήριξη, για τη στήριξη ρευστότητας και τη μείωση ίσπραξη φόρων. Όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό, τον τακτικό προπολογισμό. Και πρέπει να διατηρηθεί η τακτική κανονική δημοσιονομική πειθαρχία. Πότε ξεκινάει η ανάκαμψη, από ποια χρονική στιγμή. Όταν κρίνουμε ότι έχουμε θέσει έλεγχο τον ιό, τότε ξεκινά. Ότι δηλαδή ο κίνδυνος να υπάρξει κατάρρευση συστήματος υγείας και νέα απομόνωση νέος περιορισμός, εγκλισμός. Αυτός, αυτή είναι η ε, στιγμή. Αν είναι τόσο ε, χαμηλά αυτά τα επίπεδα ανησυχίας και κινδύνου, τότε μπορεί να ξεκινήσει κανείς ε, να περνά στην αποκράση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκαμπόρ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν θέλω να πω σε θέματα νομιμότητας και αναλογικότητας. Αυτά θα τα απαντήσει η Bundesbank. Αλλά σε ό,τι αφορά την προσωπική μου άποψη, που έχω μελετήσει την νομισματική πολιτική, νομισματική ιστορία, νομίζω ότι η ΕΚΤΑ ε, έχει σημαντικά ε, μέτρα να λεπόψει για τη μετάδοση νομισματικής πολιτικής. Εγώ μιλούσα για τους ιδρυτές Είπα ότι δεν έλαβαν υπόψη τις αλλαγέ που θα συντελούνταν σύν το χρόνο. Και αν μελετήσει κάποιο τη νομισματική ιστορία, βλέπει ότι αλλάζουν οι χρηματοπιστωτικέ δομέ και η ιδιωτική χρηματοδότηση, τα ιδιωτικά οικονομικά και οι θεσμοί ε, μακροοικονομικής πολιτικής χάνουν την αποτελεσματικότητά τους αν δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές στα ε, οικονομικά. Βλέπουμε ότι είναι η σπονδυλική στήλη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κρατικό μόλγα. Το αναγνωρίζει αυτό η έκτοτη το κόστος ε, κρατικού δανεισμού ανέβει, τότε το κόστος ε, δημιουργίας ιδιωτικής πίστης ε, ανεβαίνει. Και αν θέλουμε να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός μετάδοσης, θα πρέπει να γίνει μέσω των αγορών κρατικών ομολόγων, γιατί δεν υπάρχουν άλλα πλασματικά εργαλεία Κατά την άποψή μου, ήδη αυτή είναι μια δομική αλλαγή που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε με δημοκρατικό τρόπο ε, τον ανάγκη συντονισμού δημοσιονομικής νομισματικής πολιτικής. Έχουμε δημοκρατικούς τρόπους για να συζητήσουμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο γίνεται αυτός ο συντονισμός. Σέβομαι βέβαια και συμφωνώ με την έκτη και τη δράση της, αλλά νομίζω ότι η δημοκρατικά εκλεγμένη πολιτική είναι αυτή που θα πρέπει να έχουν επίσης λόγο για τους τρόπους με τους οποίους οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν μη συμβατικά μέτρα. Τα λέω μη συμβατικά πολύ απλά γιατί το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής που έχουμε έχει κατά κάποιο τρόπο ξεπεραστεί. Θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε νέους τρόπους, νέους ε, μηχανισμούς συντονισμού και αν απαιτείται αλλαγή των συνθήκων εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ ενός τέτοιου βήματος. Αυτό το οποίο μου προκαλεί ανησυχία και το βλέπω και στη συζήτηση που έχουμε σήμερα, ότι υπάρχει το θέμα της αλληλουχίας, ε, δηλαδή τι βάζουμε πρώτα και τι βάζουμε μετά, την ε, ανάπτυξη, τη βασιμότητα του χρέους ε, ή τούμπαλιν και αν δώσουμε προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση ή τη βιωσιμότητα, ανάλογα με το τι επιλέξουμε, κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει με την ε, χρήση των εργαλείων της μακροοικονομικής πολιτικής που έχει εκτός Ευρωζώνης. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στον τρίτο γύρο. Έχουμε τρεις ε, ομιλητές από τους πράσινους, του κύριο Κλωτ Κρουφά. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Με ακούτε? Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που αφιερώνουμε χρόνο σε αυτές τις πολύ επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων. Έχω κάποιες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά α, τους επιχειρηματίες, μιας και είμαι επιχειρηματίας. Ε, αναρωτιέμαι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, τα αριθμητικά, τα ποσά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εργαλείο Next Generation. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία από πού προέρχονται και πώς μπορούν να οριστούν σαν τέτοιο κείμενο. Η κυρία Φαντερ Λάιεν μίλησε για 500 εκατομμύρια. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τα δισεκατομμύρια. Πώς μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε αυτό το ποσό. Πώς θα ξέρουμε αν ε, δεν ε, θα αλλάξει το ποσό αυτό ανάλογα και με τις εξελίξεις και τις οικονομικές ε, εξελίξεις στην αγορά. Για να εκτιμήσουμε λοιπόν τον πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο ε, και να μην ε, καταργηθούν οι οικονομίες μας. Η οικονομία προφανώς δεν είναι ακριβής επιστήμη, είναι ε, κοινωνική επιστήμη και ίσως τα 40 τελευταία χρόνια μας έχουν κάνει να το ξεχάσουμε αυτό. Αν είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια πραγματική οικονομία, μια οικονομία κοινωνική, θα πρέπει να εξυπηρετούμε τον άνθρωπο. Αυτό θα μπορούσε να αναφερθεί στις πολιτικές εκθέσεις και τις πολιτικές ε, Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αυτή η διάσταση δηλαδή η πραγματική, της πραγματικής οικονομίας. Προκειμένου να εξέλθουμε λοιπόν από την κρίση, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στις επιχειρήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το ίδια με, με αυτή που ήταν πριν. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν κάποια μοντέλα οικονομικής δραστηριότητας έχουν επιβιώσει με πιο στεναρό τρόπο της κρίσης. Κυρίως, για παράδειγμα, τους συνεταιρισμούς. Ε, πρόκειται για ε, ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο ενδεχομένω να μας είναι χρήσιμο. Και έτσι Βλέπουμε ότι σε όλο τον 20ο αιώνα με τον τρόπο αυτό ε, ολόκληρε επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει στον ε, τομέα για παράδειγμα της, ε, των τη της αλίας, ακόμα και για τις τράπεζες. Κύριε Γκριφά, θα μπορούσατε παρακαλώ να κάνετε τα καταληκτικά σας σχόλια, σχόλια λέει ο Πρόεδρος. Ναι. Όταν λοιπόν δίνουμε τέτοιες μεγάλες υποστηρίξεις ε, και τόσο μεγάλα κεφαλικές ενέσεις ε, δεν θα μπορούσαμε παράλληλα να προτείνουμε να δώσουμε και στους ε, εργαζόμενους που το επιθυμούν το κεφάλαιο που χρειάζονται για να μπορέσουν να διχρηστούν τις επιχειρήσεις τους. Για να είμαστε λοιπόν σε επίπεδο κοινωνικής οικονομίας. Ναι, θα πρέπει να κάνετε τα καταλητικά σας σχόλια, κύριε Γρυφά, λέει ο πρόεδρος. Έχετε λοιπόν αριθμητικά στοιχεία για τον αντίκτυπο της κρίσης σε ό,τι αφορά το μοντέλο των συνεταιρισμών και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να έχουν πιο ανθεκτική πορεία τέτοιε επιχειρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κρυφά, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα, τον κύριο Έπινγκ. Μα δεν είναι το λόγο στον εαυτό μου, το συνονόματό μου. Να ρωτήσω λοιπόν μία ερώτηση και έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο Χοχντάν. Μιλήσατε για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και λέμε ότι ενδεχομένως, μάλλον το Μάιο, τα χαμηλά επιτόκια και το καθεστώς ε, με επικέντρωση στο χρέος ενδεχομένω να ε, αποτρέψει την ΕΚΤΑ από την άσκηση της εντολής της και θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής, του ευρώ και των κρατών μέλλον. Πιστεύετε λοιπόν ότι το ευρώ θα βγει εκτός ελέγχου και ποιο είναι το δεύτερο σχέδιο αν συμβεί κάτι τέτοιο και κατά δεύτερον πώς εκτιμάτε το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα συνεχίζω με τον εκπρόσωπο της ΓΚΟΕ, τον κύριο Μάικ Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Για τον κύριο Γκουρίτσια, καταρχά, η πρώτη μου ερώτηση μα είπατε ότι από το 12% των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και ότι δεν μπορούμε να σώσουμε όλε τι επιχειρήσει, αλλά παράλληλα φοβάστε ότι δεν θα βοηθήσουμε τι μικρέ επιχειρήσει. Πώ λοιπόν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτό για να εξασφαλίσουμε ότι θα πάρουν επαρκή υποστήριξη αυτέ οι επιχειρήσει οι μικρέ. Και επειδή οι πιο πολλέ τράπεζε στην Ευρώπη είναι ιδιωτικέ, πολλέ ε, δεν ε, διατίθενται ετιτέρως να υποστηρίξουν μικρέ ε, επιχειρήσει Χρειάζεται κρατική λοιπόν υποστήριξη. και σε ό,τι αφορά τη χαλάρωση των δημοσιονομικών ε, κανόνων. Πιστεύετε ότι οι κανόνε αυτοί θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να βοηθήσουν τι μικρέ επιχειρήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μια δεύτερη ερώτηση προ την Δανιέλα. Διανέλια, Δανιέλα, αναρωτιέμαι. Πιστεύετε ότι έχει ξεπεράσει το οικονομικό μα σύστημα με τον Bretton Woods ε, τη δεκαετία του 40 μειώθηκαν ε, το βιωτικό επίπεδο και από την ε, πτώση του Bretton Woods και μετά το Ρίγκαν το 1971. Τώρα, πιστεύετε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λογική του νέου φιλελευθερισμού κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, ουσιαστικά την αφήνουμε κατά μέρος. Χρειάζονται συλλογική αλληλεγγύη σε περιπτώσει κρίσης για να υποστηρίξουμε τη συλλογική ευημερία. Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε προτού επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κουρίνσας για να απαντήσει στις ερωτήσεις που του ετέθησαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Να σας απαντήσω καταρχάς για το μέγεθος, το όγκο του Next Generation. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να μην αναρωτηθούμε κατά πόσο θα αρκέσει το ποσό του Next Generation. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να τονίσουμε όμως ότι πρόκειται για ένα καινούργιο εργαλείο. Δεν είναι εντελώ καινούργιο γιατί από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης υπήρχε ιδέα. Ακόμα και από τον Μάντελ δεκαετία του που έλεγαν ότι αν υπάρχει μια οικονομική ένωση θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη για μεγάλα σύμμετρα σοκ. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο κλειδονισμό τώρα. Έχουμε και ένα δεύτερο. Είχαμε μάλλον ένα πρώτο τέτοιο σοκ με την χρηματοοικονομική κρίση. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο τέτοιο σοκ με την πανδημία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε το οικονομικό σύστημα στο σύνολό του να μην καταρρεύσει και να πάρει μαζί του και όλα τα κράτη. Στην περίπτωση της πανδημίας χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια αμοιβαία υποστήριξη και είναι σημαντική η υποστήριξη το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο πλέον και ότι υπολογίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το εργαλείο αυτό και να επιβιώσει και να ανακάμψει στις διεθνείς αγορές και να υπάρξει αμοιβαιοποίηση κάποιων τέτοιων συστημάτων. Δεν με απασχολεί κατά πόσο να αρκεί το ποσό αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αρκέσει, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη στην παρούσα φάση τελειωτική. Δεύτερη ερώτηση. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το νέο μοντέλο. Κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Φυσικά, σε έναν βαθμό ναι. Αλλά να είμαστε και ξεκάθαροι. Η αρχή ότι υπάρχει ένας στόχος για κάθε, κάθε πολιτική μάλλον όπως ένα στόχο εξακολουθεί να ισχύει. Αν θέλουμε να κοιτάξουμε λοιπόν την πράσινη πολιτική και άλλους ε, στόχους και το πώς θέλουμε να πετύχουμε επιθυμητικούς στόχους, θα πρέπει να δούμε, να μην ε, χρησιμοποιήσουμε τα ίδια εργαλεία για τους ίδιους στόχους. Θα θέλαμε λοιπόν να, να διαμορφώσουμε τις, τα θεσμικά όργανα μπορεί να μην σκεφτόμαστε αρκετά ευρέως για το πώς θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό καλά θα κάνουμε να το έχουμε υπόψη μας, θεωρώ. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χόκταν για τις ερωτήσεις που του έκανα. Μία ερώτηση του έκανα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ και με χαρά να απαντήσω στα δύο σκέλη της ερώτησης για την ανάκαμψη, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω κάποια ερωτηματικά εδώ σε ό,τι αφορά ένα ταμείο για το θέμα αυτό. Καταρχάς, δεν καλύπτει το θέμα των κενών και των αποθεματικών τα οποία ανέφερα και στην ομιλία μου. Ούτε σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του κορονοϊού αρκεί στις διάφορες χώρες, στην τρέχουσα μορφή. Και δεν υπάρχει επαρκής αιρεσιμότητα, θεωρώ, για το ποιος παίρνει χρήματα. Αυτό οδηγεί σε μεγάλες δαπάνες, μεγάλους φόρους. Μία εναλλακτική θα μπορούσε να είναι να δημιουργηθούν όροι υπό τους οποίους θα μπορέσουν να ανθίσουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και κοιτώντας τέλος ε, το σκέλος των δαπανών και βλέπουμε ότι πολλά χρήματα πηγαίνουν στο Green Deal, στην Πράσινη Συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την, ε, το προσέγγισμα της οικονομίας είναι καλό, αλλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και να προσέξουμε, γιατί δεν θέλουμε επίσης να περάσουμε σε μέτρα προστατευτισμού και σε ό,τι αφορά την ατζέντα ψηφιοποίησης να κοιτάξουμε, μην πέσουμε στην παγίδα του να προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τους νικητές για το... στην επόμενη περίοδο. Να δημιουργηθούν λοιπόν συνθήκες ανάπτυξης παρά να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη. Για, για το ευρώ, το οποίο ενδεχομένω να ξεφύγει από τον έλεγχο. Τα χαμηλά και θεωρώ ότι θα είναι μη βιώσιμα σε μεγάλο βάθο χρόνο. Η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα πιστοτικής χαλάρωσης ή, εν πάση περιπτώσει, ότι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει πληθωρισμό και αστάθεια. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Τι θα πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα για την ανάκαμψη της βιωσιμότητας και για την ανάκαμψη των buffer αυτών των αποθεμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα σύγκληση θα έλεγα στην Ευρωζώνη αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορα πλαίσια. Δεν νομίζω ότι το τρέχον πλαίσιο, νομίζω μάλλον ότι το τρέχον πλαίσιο φτάνει στα όρια του. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών στην Ευρωζώνη. Για να βρεθούν νέοι κοινοί τόποι και αυτό προφανώς θα εξαρτηθεί και από τις πολιτικές προτιμήσεις. Μπορούμε να κινηθούμε πιο, με πιο πολύ διαφάνεια προς την κατεύθυνση μιας δημοσιονομικής ε, ένωσης ή πολιτικής ένωσης, ε, ενδεχομένω ανάλογα με τις πολιτικές ε, του καθενός. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να κινηθούμε και προς μια πιο ευέλικτη ευρωζώνη. Αυτό θα ήταν ένα δεύτερο σενάριο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Και τέλος και η κυρία Γκαμπόρ για να απαντήσει στα ερωτήματα που τη ετέθησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εν συντομία, νομίζω ότι συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητέ ότι δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος για να καταλήξουμε για τα 500 δι ε, σε, ε, και τα 50 δις επιπλέον. Αλλά υπάρχουν τα πολιτικά αμα, δείγματα που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε φάση που θα μπορούσε να δεχτεί μια υπερεθνική οικονομική δύναμη. για να υπάρξει ανάκαμψη δεδομένης και της ευάλωτης θέσης. Και αυτό εξαρτάται και από τη Γερμανία και τα τεράστια πλανεκτήματα που έχει για να ορίσει τα ασφαλή αποθέματα, Γιατί το κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπιζόμαστε και να προσπιζόμαστε τον νέο φιλελευθερισμό. Θεωρώ ότι ζούμε ακόμα σε μια εποχή παγκοσμιοποίηση. Δεν έχει μεταρρυθμιστεί ακόμα ε, παρκώς ο χρηματοοικονομικός κλάδος. Δεν, χρειάζεται να υποθυμίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έγινε το 2008 και όλες οι προσπάθειες που έγιναν μετά με την προσπάθεια φορολόγησης ε, των συναλλαγών για να υπάρξει αλληλοεξάρτηση σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέο των χωρών. Χρειάζεται λοιπόν, ε, αν δεν υπάρξουν οι αλλαγές αυτές, ε, χρειάζεται αντιάρθρωση των ε, ιδιωτικών κλάδων και ίσως να υπάρξει δυνατότητα να αναβιωθεί αυτό τόσο ο να συναλλαγών υπός πράσινης μορφή ενδεχομένω για να μπορέσει να τονωθεί και να υποστηριχθεί η οικονομική ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Σίγουρα οι ευρωβουλευτές της ΕΚΟΝ θα λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις σας σε οποιαδήποτε απάντηση και πρωτοβουλία αναλυφθεί στο μέλλον. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά για να ελέγξουμε τις συνδέσεις με τους επόμενους ομιλητές που έχουμε στο δεύτερο πάνελ μας. Good afternoon, Mrs. This is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 για την πολιτική ανταπόκριση στην πανδημία COVID-19 συμπεριλαμβανομένων νομισματικών και δημοσιονομικών μέτρων. Έχουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες. Καλωσορίζουμε δύο επικεφαλής οικονομολόγους. Ο ένας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η κυρία Τζίτα Κόπινατ και η δεύτερη είναι από τον ΟΣΑ, η κυρία Λοράνς Μπον. Έχουμε επίσης τον κύριο Βλαντιμίρο Τζακέ, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών στη Ρώμη και τέλος την κυρία Αν Πέτιφορ, που είναι ε, πολιτική οικονομολόγος, συγγραφέας πολλών ε, βιβλίων σχετικά με την ε, κρίση και την απάντηση σε αυτή. Καλώς ήρθατε όλοι στην Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα θα δώσω όμως το λόγο στην Πρόεδρό μας, την κυρία Τινάλη, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους προηγούμενους εμπειρογνώμονες για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και καλωσορίσω και τους επόμενους ομιλητές μας που είναι εξέχουσες προσωπικότητες. Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο να έρθετε και να συμμετάσχετε. Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να έχει τέτοιου είδους διάλογο με τους ε, κύριους παίκτες, με τους εμπειρογνώμονες. Ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές ότι ζούμε σε περίοδο αβεβαιότητας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς με ακρίβεια προγνωστικά. Αυτό όμω που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι να αναλύσουμε και να μάθουμε από το παρελθόν, να καταλάβουμε καλύτερα από τα λάθη μας τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, τι άλλα πεδία θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε. Όλα αυτά μας βεθούν πάρα πολύ για να καταλήξουμε στις σωστές αποφάσεις πολιτικής και μέτρων. Έτσι ευρύνονται οι προοπτικές μας και καταλαβαίνουμε καλύτερα ποια είναι η κατάσταση. Οι επόμενοι ομιλητές σίγουρα θα μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση με τις γνώσεις τους. Και πάλι ευχαριστώ πολύ την κυρία Κόπινα, την κυρία Μπον, τον κύριο Τζακέ και την κυρία Πέτιφορ ελπίζω σύντομα να μπορέσω να σας υποδεχτώ και στις Βρυξέλλες διαζώσεις. Τον Ιούλιο ήταν να πάω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον, αλλά δυστυχώ χρειάστηκε να κυρώσω το ταξίδι αυτό. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Ο κύριος Σέπινγκ, ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασής μας που πρόκειται για την ανταπόκριση στην κρίση COVID-19 συμπεριλαμβανομένων μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για να έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το έργο των νομοθετών μας. Έχουμε οργανώσει τη διεξαγωγή της ακρόασης αυτή ως εξή. Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις θα ξεκινήσω γύρω των ε, παρεμβάσεων 7 λεπτά για τον κάθε ομιλητή εμπειρογνώμονα. Μετά θα έχουμε γύρους ε, ερωταπαντήσεων με δύο ή τρεις ερωτήσεις κάθε φορά και παρατηρήσεις στο τέλος από την Πρόεδρο. Για άλλη μια φορά σας ζητώ να τηρείτε το χρόνο σας. Τέλος, για τη διερμηνία. Έχουμε διερμηνία για τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα πολωνικά. Και αυτό μέχρι τις 17 και 45, μέχρι τις 6 παρατέταρτο θα έχουμε διερμηνία. Μετά θα συνεχίσουμε στα αγγλικά μόνο. Τώρα λοιπόν, το λόγο έχουν για 7 λεπτά οι ομιλητές μας και αρχίζουμε με την κυρία Τζίτα Κοπινάτ, που είναι επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με προσκαλέσατε να έρθω να σας μιλήσω για την ανταπόκριση στην κρίση του κορονοϊού. Έχουν περάσει τρεις μήνες από το ξέσπασμα της πανδημίας, κάτι το οποίο οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε μια κρίση ανευπροηγουμένου το μέγεθος της κρίσης αυτής, ο μεγάλος εγκλισμός όπως θα τον έλεγα, είναι πραγματικά χωρίς προηγούμενο από την μεγάλη ύφεση τόσο για τις προηγμένες οικονομίες όσο και για τις αναδιόμενες αγορές που φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε ύφεση συγχρόνως. Καμία χώρα, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στον κόσμο δεν έχει γλιτώσει τις κοινωνικές, οικονομικές συνέπειες και τις συνέπειες στον τομέα της υγείας. Η Ευρώπη ήταν μία από τις πρώτες περιοχές του κόσμου που επλήγει από την ε, πανδημία. Η ανάκαμψη φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πιο μεγάλη και περισσότερο ενισχυμένη από ό,τι περιμέναμε τον Απρίλιο. Και ακόμα και όταν θα έρθει η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρόλα αυτά ε, θα παραμείνουν τα αποτελέσματα χαμηλότερα από το βαθμό που είχαμε πριν από την κρίση με διαρθρωτική ανεργία και χαμηλή παραγωγικότητα. Η πολιτική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν στην κρίση κρίνεται από την ταχύτητα, το μέγεθος και το βάθος. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε βγει από τις δυσκολίε και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ένα δεύτερο κύμα ε, κορονοϊού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τώρα να προσέξουμε τι πολιτικές χρειάζονται για να στηρίξουμε μια ισχυρή ανάκαμψη και να αποφύγουμε μόνιμες σουλές από την κρίση αυτή. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, τη απουσία ιατρικής λύσης το να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος στην υγεία παραμένει προτερότητα. Οι χώρες θα πρέπει να προσαρμόσουν ε, τις παρεμβάσεις τους ανάλογα με την κατάσταση. Αλλά ε, γενικά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ένα ικανοποιητικό σύστημα υγείας με ικανότητα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και οι πρακτικές ε, τήρησης κοινωνικών αποστάσεων όπως επίσης και άλλοι περιορισμοί από τη μία και από την άλλη μεριά να ελαχιστοποιήσουμε τις οικονομικές διαταραχές. Οι πολιτικές χρειάζονται τώρα για να διασφαλίσουν επίσης την κατάλληλη παραγωγή και την διανομή εμβολίων. Μια δεύτερη προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους με μέτρα που είναι για παράδειγμα η προσωρινή απασχόληση, η αποφυγή απολύσεων. Κίνδυνοι υπάρχουν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας όπως είναι η φιλοξενία, τα ταξίδια που θα δυσκολευτούν να κερδίσουν πάλι τη ζήτηση που είχαν κατά το παρελθόν και θα υπάρχει η επιβράδυνση για καιρό ακόμα μετά την κρίση. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, λοιπόν, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν σε διάφορα μέτωπα. Πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τους εργαζόμενους με καλά σχεδιασμένα προγράμματα προσωρινής απασχόλησης και να διευκολύνουν επίσης και την ανακατανομή τους σε κλάδους όπου οι προοπτικές για ανάπτυξη είναι καλύτερε. Οι πολιτικέ αυτέ μπορούν να βοηθήσουν εφόσον συμπεριλαμβάνουν και ενίσχυση των μισθών, επιδοτήσει, επανακατάρτιση κλπ. Η ευρωπαϊκή αγορά ε, εργασίας περιλαμβάνει τις συλλογικέ συμβάσεις, την προστασία της απασχόλησης, ε, συστήματα ενίσχυσης και επιδομάτων και αυτά πρέπει να παραμείνουν. Μια τρίτη πολιτική προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίοι βρίσκονται σε πρόβλημα δεν θα καταλήξουν σε πτώχευση. Οι κυβερνήσεις πρέπει να περάσουν από την ανησυχία που έχουν για την ρευστότητα σε μια διαδικασία ελαχιστοποίησης των πτωχεύσεων. Τώρα υπάρχουν διάφορα δίκτυα και διασυνοριακά στην Ευρώπη, σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με συντονισμό για να διευκολυνθεί η συνέχιση δραστηριότητας των επιχειρήσεων και η ανακατανομή των ε, πόρων από τις μη φερέγγες επιχειρήσεις της φερέγγες. Αυτός ο μεγάλος εγκλισμός έχει επίσης ενισχύσει τη φτώχεια και τις ανισότητες. Σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα πράγματα και οι πολιτικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα βελτιώσουμε τα συστήματα κοινωνικής ε, πρόνοιας, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, για την ζωτική σημασία για την επεκατανομή των δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Η μεγάλη αβεβαιότητα στο δρόμο προς την ε, ανάκαμψη ε, οφείλεται στο ότι δεν γνωρίζουμε καλά πώς θα προχωρήσει η πανδημία. Πρέπει όμως να υπάρξει εκ νέου εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη στις επιμέρους χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που πρέπει να δράσουν συντονισμένα. Το στάδιο της ανάκαμψης αποτελεί και μια ευκαιρία για μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο χρέος μετά την κρίση. Χρειάζονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις ε, για να ενισχυθεί η ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης και μετά. Κάποιε χώρε επιτέλεσαν πρόοδο βέβαια τα τελευταία χρόνια. Χρειάζονται όμω περισσότερα πράγματα όσον αφορά μεταρρυθμίσει στον εργασιακό τομέα και στην παραγωγή. Επιπλέον, έχουμε μπροστά μα και μια ευκαιρία για να επιταχύνουμε και το πρασίνισμα των οικονομιών μα και την ε, ψηφιακή μετάβαση. Κάποιε χώρε έχουν θέσει φιλόδοξου στόχου, αλλά χρειάζονται περισσότερε δράσει ευρύτερα. Μετά λοιπόν την παγκόσμια οικονομική κρίση δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και δημιουργήθηκε επίσης η Τραπεζική Ένωση και έγιναν πολλά βήματα για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Νομισματική Ένωση για να ενισχυθεί η αντοχή, να συμπληρωθεί η Τραπεζική Ένωση ή να έχουμε μια πιο ισχυρή κεφαλαιακή αγορά κλπ. Τώρα θα ολοκληρώσω λέγοντας τα Η πρόταση Next Generation EU που ακούσαμε τον Μάιο αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια για συνεργασία στην οικονομική πολιτική που θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για μια ισχυρή ευρωπαϊκή ανάκαμψη και συγχρόνως να ενισχύσει την αντίληψη των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά την συνοχή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ε, Νομισματικής Ένωσης, που μαζί μπορούν ε, να ενισχύσουν και το ρόλο του ευρώ ως διεθνές νόμισμα. Τέλος, η κρίση αυτή θέτει και το θέμα των ε, κινδύνων στους οποίους μπορεί να οδηγηθούμε με ενίσχυση του προστατευτισμού. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει τα πάντα για να το αποφύγει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε την κυρία Λόρανς Μπούνα, που είναι επικεφαλής οικονομολόγος στον ΟΣΑ. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως γνωρίζετε, ΣΑ μόλις δημοσίευσε τις αρινές οικονομικές προοπτικές για το 2020 με τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, έκτακτη και διάχυτη καθολική αβεβαιότητα, έκτακτους κραδασμούς ε, και έκτακτη ανταπόκριση με συγκεκριμένε πολιτικέ και επίση έκτακτη ευρωπαϊκή ανταπόκριση. Και θα ήθελα να εστιάσω εδώ τι παρατηρήσει μου κυρίω στον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή ανταπόκριση θα ε, είναι επαρκή ε, για να αντιμετωπίσει τι όλο και ογκούμενε ε, αποκλήσει που προκύπτουν στην Ευρώπη λόγω τη κρίση. Ό,τι αφορά την αβεβαιότητα, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, διότι ίσω σημαίνει ότι πρέπει κάποια πράγματα να εφαρμοστούν διαφορετικά ή κάποια περισσότερα πράγματα θα πρέπει να γίνουν πιο, το πιο αβέβαιο είναι πια, θα είναι η προοπτική της επιδημίας και αυτό θα επηρεάσει και τις οικονομικές προοπτικές. Δεν θα έχουμε ένα εμβόλιο ε, ή μια θεραπεία για τους επόμενους 12 ή 18 μήνες ε, τουλάχιστον που σημαίνει ότι τα μέτρα τήρηση αποστάσεων, ε, οι κανονισμοί υγείας, υγιεινής θα είναι μαζί μας για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα οδηγώντας σε αύξηση κόστου σε διάφορες τομείς και σίγουρα θα επηρεάσουν δομικά τις ε, δράσεις στην οικονομία. Επίσης ε, δεν θα ανοίξουν όλα τα σύνορα ε, ακριβώς όπως πριν. Και για μεγάλες χρονικές ε, περιόδους θα, θα υποστούν ζημία κάποιοι τομείς, θα χρειαστεί να υπάρξουν δομικές αλλαγές για οικονομίες, άλλοι τομείς μπορεί να ανθίσουν και όλα αυτά επηρεάζουν και την αγορά και, την, ε, και το κεφάλαιο. Επίσης μπορεί να προκύψει και νέα έξαρση της επιδημίας, ε, αν όχι σε παγκόσμιο πέδο, σε περιφερειακό, κάποιοι δηλαδή μπορεί να χρειάζεται πάλι να απομονωθούν είτε τομείς είτε κατηγορίες πληθυσμού και επομένως χρειάζεται Ενδεχομένω να έχουν υπόψη ότι θα χρειαστεί στο μέλλον υποστήριξη. Πρέπει λοιπόν η οικονομική πολιτική πρώτα απ' όλα να προσπαθήσει να μειώσει αυτή την ανασφάλεια. Το δεύτερο είναι οι έκτακτοι κραδασμοί και οι δημόσιε παρεμβάσει. Ξέρετε ότι οι οικονομικέ δραστηριότητε κατέρευσαν ε, με τι ε, με, με τα μέτρα απομόνωσης ε, και το κλείσιμο επιχειρήσεων ε, στις χώρες του ΩΣΑ, σε κάποιες χώρες από 20 έως 30% και προβλέπουμε στην παγκόσμια οικονομία συρρήκνωση 6 έως 7,5 μονάδων 6 ε, 7,5% φέτος και για την Ευρωζώνη 9 με 11,5%. Επίσης η ανάκαμψη θα είναι περιορισμένη και έτσι θα έχουμε απόλυση οδήματος κατά κεφαλή γύρω στο 10% με διακοιμάσεις ανάλογα με τις χώρες. Οι ευρωπαϊκές χώρες αντέχουν αντέδρασαν γρήγορα στις οικονομικές αυτές, ε, στους οικονομικούς αυτούς κραδασμούς, πρώτα σε εθνικό και μετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερες δράσανε ανελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο για τη στήριξη των συστημάτων υγείας, των εργαζομένων και την υιοθέτηση ε, σχεδίων βραχυπρόθεσμης απασχόλησης και μέσω κάποιων εγγυήσεων, δανείων και αναστολής ε, καταβολής φόρων και η ειδική υποστήριξη δίνεται σε κάποιου τομεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε πιο γρήγορη και ευρύ αντιμετώπιση και η Κομισιόν πολύ γρήγορα ήρε κανόνες δημοσιονομικού κρατικών ενισχύσεων που θα επηρέαζαν και θα περιόριζαν την εθνική ανταπόκριση. Επίση, έχουμε διάφορους διάφορα προγράμματα στοχευμένα, το ΣΟΥΡ, το, τις ε, διευκολύνσεις της ΕΤΕΠ, ε, το πρόγραμμα πανδημίας ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και το Ταμείο Ανάκτησης, Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η έκτεπη αντέδρασε γρήγορα και έγκαιρα, είχε και ε, αυτό το πρόγραμμα ε, προωθήσει για την αγορά στοιχείων ενεργητικού τομέα στι δευτερογενεί αγορέ, ε, που είναι σημαντικό και Σίγουρα δίνουν όλα αυτά τα προγράμματα μήνυμα αισιοδοξία και είναι πολύ σημαντικό γιατί η Εθνική Δημοσιονομική Υποστήριξη μαζί με το βάθο τη ύφεση το δημόσιο χρέο ε, θα το εκτινάξει ε, κατά 20 ποσοστέ ε, μονάδε στην Ένωση. Και αυτή η αύξηση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί στήριξη και για το δεύτερο εξάμεινο του 20 και για το 2021. Πολλά θα εξαρτηθούν δε από την ταχύτητα τη ανάκαμψη και από το πόσο ε, θα επιτύχει αυτή η υποστήριξη. Είναι αρκετή. Πρώτα απ' όλα, τα πακέτα, ε, τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά, ίσως χρειαστεί να αυξηθούν σε μέγεθος. Ε, οι οικονομικές μας προοπτικές δείχνουν ότι το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη θα εξακολουθήσει να είναι 7 κάτω των ποσοστών του 2019 με το τέλη του 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα προγράμματα και σχέδια. Άρα φαίνεται ότι μπορεί ε, να υπάρξει ανάγκη για πιο ενισχυμένη και συντονισμένη υποστήριξη. Και αυτό έχει να κάνει με τις εθνικές χώρες. Ε, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η, η αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων να παραμείνει αναλύτω και το 2021 που θα χρειαστεί μεγαλύτερο προπολογισμό για την ανάκαμψη. Επίση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει το χρονοδιάγραμμα για το ταμείο αυτό τη ε, ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Δεν θα υπάρχουν πολλά ε, κεφάλαια διαθέσιμα στην περίοδο 2020-2021 και ότι ο μεγαλύτερο, τα μεγαλύτερα κίνητα θα δοθούν και ερευνούν το 2023-2024. Θα... Είναι πολύ αργά αυτό για πολλέ επιχειρήσει και πολλέ οικογένειε. Επομένως, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γρήγορα να τεθεί σε εφαρμογή. Και το θέμα επίση που προκύπτει είναι εάν μπορεί να γίνει μια εμπροστοβαρή χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. Γιατί αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, απτόχευσης, αφαιρεγγιότητας και αν θέλουμε να μην πέσει σε βαθιά κρίση, με ακόμα πιο βαθιά η ευρωπαϊκή οικονομία, θα χρειαστεί δημόσια υποστήριξη στο δεύτερο εξάμενο του έτους και το 2021 κυρίω. Επίσης, ε, η COVID-21 οδήγησε σε ασύμετρους κραδασμούς σε όλο τον πλανήτη, αλλά ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως γνωρίζετε, οι οικονομικές επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με τους ε, παράγοντες του υγειονομικούς, ε, κάποια τοπικά στοιχεία όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού ή η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, από οικονομικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται όπως είναι εξειδίκευση ανατομέα ή η βιομηχανική δομή και διάρθρωση, το μέγεθος δηλαδή των επιχειρήσεων που συγκροτούν τον ιστό ε, της οικονομίας. Ε, και ίσως έτσι υπάρξει όξυνση των αποκλήσεων και διαφορών ε, μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Μέχρι τα τέλη του 2021, για παράδειγμα, το ΑΕΠ κατά κεφαλή στην Ισπανία θα μπορούσε να είναι περισσότερο από 35% χαμηλότερο από ό,τι της Γερμανίας, της Ιταλίας 30% και της Ολλανδίας 12% πάνω από 12% παραπάνω. Και υπάρχει μια κλίδα κατανομής που προκύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχει ένα στοιχείο ανακατανομής από το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτιμότητας, αλλά στο βαθμό που αυτό το στοιχείο της ανακατανομής στοχεύει σε τομείς και χώρες που πλήττονται περισσότερο, ε, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό ε, θα υπάρχει αυτό, ε, θα επηρεάσει αυτή η κλίδα ανακατανομής Και όλα θα εξαρτηθούν βέβαια και από το πόσο σημαντική είναι αυτή η οικονομική ε, κράτηση και το οικονομικό σόκα ανάλογα με τη χώρα. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουν αρθεί οι κανόνε ε, περί κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι καλοδεχούμενο. Όμω αυτέ οι παρεμβάσει είναι σημαντικέ όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ποσότητα αλλά και την ποιότητά του. Και μέχρι στιγμή υπάρχει μεγάλη διαφορά, διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά ε, τι ενισχύσει και το πώ χρησιμοποιούνται. Κάποιε ε, χώρε στηρίζουν τι επιχειρήσει του κυρίω με εγγύσει δανείων, ενώ άλλε με εισοδηματική, με κεφαλιακή υποστήριξη. Μπαίνουμε σε μια φάση τώρα που οι κυβερνήσει μπορεί να μειώσουν ε, την υποστήριξη που, άρχισα, που έδιναν στην πρώτη φάση και να υπάρξει ζήτημα επιστοτική επιφάνειας για πολλές επιχειρήσεις. Ε, και οι επιχειρήσεις που έλαβαν ε, εισοδηματική υποστήριξη, που πήραν κάποια κονδύλια, κάποια κεφάλαια, μάλλον θα είναι πιο ανθεκτικές, ενώ εκεί που υπήρξαν περισσότερα δάνεια, η εγγύηση δανείων, η φερεγγιότητα των επιχειρήσεων μπορεί να επιδεινωθεί και να έχουμε χρεοκοπίες και αύξηση του δημόσιου χρέους. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η ευρωπαϊκή απάντηση δεν είναι επαρκής όσο δεν έχουμε ένα, ε, ένα εργαλείο σταθεροποίησης. Χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο. Ε, και τη σταθεροποίηση μέχρι στιγμή την έχει αναλάβει μόνο η έκταρα. Εδώ λείπει ένα σκέλος ε, της πολιτικής. Ευχαριστώ. Βλατιμίρο Τζακέ, από τη Ρώμη, ο επόμενο ομιλητής. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ευρύ θα επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, στον τραπεζικό κλάδο. Και διάλεξα το θέμα αυτό για δύο λόγους. Όπως είπε η EBA σε ένα πρόσφατο έγγραφο, η ποιότητα των οικονομικών στοιχείων αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες λόγω πιθανής αύξησης, προφανής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και παράλληλα ξέρουμε ότι η διαδικασία διαδανεισμού είναι κρίσιμος παράγοντας για να μπορέσει να υπάρξει γρήγορα οικονομική ανάκαμψη. Γνωρίζουν λοιπόν οι πολιτικοί την στρατηγική σημασία του δανεισμού στο τρέχον περιβάλλον. Αντίδρασε λοιπόν γρήγορα η ΕΚΤ δίνοντας αρκετή ρευστότητα στις τράπεζες η εποπτική αρχή ε, προσωρινά χαλάρωσε κάποιες απαιτήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσείς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσαν γρήγορε λύσεις το ΣΥΡΑ 2. Πιστεύω όμως ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα τους επόμενους ε, μήνες. Δύο εξ αυτών θα αναφέρω. Προσωρινή τροποποίηση του κανονισμού 2019 630 το Απριλίου 2019 σε ό,τι αφορά την ελάχιστη κάλυψη απολειών, σε ό,τι αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, δίνοντα μια παράταση δύο ετών σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις και μια πιο ουσιώδη παράταση του νέου ορισμού της ε, αδυναμίας πληρωμής. Τέτοια μέτρα υποστηρίχτηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η ανάγκη παράταση ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, αλλά υπάρχει σοβαρός λόγος που συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι προκυκλική αυτοί οι κανόνες και εδώ λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την φιλοσοφία που υποστήριξε το κύμα ρύθμιση που επηρέασε το ευρωπαϊκό τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα μετά τη μεγάλη ύφεση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ και να σας δώσω κάποιες ε, βασικές έννοιες αυτής της φιλοσοφίας. Η επικέντρωση καταρχά είναι ο κατεξοχήν δρόμο για τον ανταγωνισμό σε παγκόσμια επίπεδο. Κατά δεύτερον, one size fits all, μία λύση για όλου. Κατά τρίτον, μεγάλη εποπτεία χρειάζονται στο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, αλλά όχι τόσο πολύ στο κίνδυνο της αγοράς. Και τέταρτον, ε, προτεραιότητα είναι η μείωση του κινδύνου. Απόλυτη προτεραιότητα. Και να σας εξηγήσω λοιπόν αυτές τις αρχές, έτσι συντομία, αν μου το επιτρέπει και ο χρόνος. Καταρχάς, το γεγονός ότι η επικέντρωση θεωρείται η καταξοχή λύση για τα θέματα ανταγωνισμού. Ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Κλάδος πέρασε μια τεράστια διαδικασία επικέντρωσης τα τελευταία χρόνια από 8.000 τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2013 σε 3.000 το 2019. Αλλά η οικονομία σε κλίμακας δεν είναι, μοναδικές, δεν είναι το μοναδικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα στην εποχή FinTech και επιπλέον να έχουμε υπόψη μας ότι κάποιες οικονομίες κλίμακας ουσιαστικά δημιουργήθηκαν από την ρύθμιση. Περνάμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη αρχή. Το δόγμα ότι μπορεί να υπάρξει μία λύση για όλους. Αν ε, απορρίψουμε οποιαδήποτε αναλογικότητα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή σύνθετων των κανονισμών, Αυτό θα αυξήσει το επίπεδο κόστος για τις μικρές τράπεζες και θα τι κάνει μη βιώσιμε. Επίσης, η τρέχουσα ρύθμιση επιτρέπει στι μεγάλες τράπεζες να χρησιμοποιήσουν λιγότερο κεφάλαιο από ότι οι πιο μικρές για τις ίδιε δραστηριότητες ε, με τα μοντέλα εσωτερική ε, αξιολόγησης. Έτσι λοιπόν ε, προωθούμε μέσω της ρύθμισης την επικέντρωση, τη συγκέντρωση τραπεζών. Τρίτο σημείο σε ό,τι αφορά την έντονη ανάγκη που υπάρχει για αποπτία του κινδύνου χρηματοδοτικού του κινδύνου και όχι τόσο πολύ του κινδύνου της αγοράς. Χρειαζόμαστε πιο πολύ κεφάλαιο από τις κεφαλαίες αγορές. Και η συνέπεια είναι ότι η χρήση του κεφαλαίου προτιμάται, ενώ η χρήση του κεφαλαίου για δανεισμό ε, δεν ε, προωθείται, αποθαρρύνεται. Εδώ να έχουμε υπόψη μας ότι καταρχάς σήμερα η μεγαλύτερη πηγή συστημικού κινδύνου για την ε, τραπεζικό κλάδο είναι το κίνδυνος από την αγορά. Όχι από τις πιστώσεις. Και δεν μπορεί οποιαδήποτε ένωση κεφαλαγορών να αποτελέσει αντικατάσταση των τραπεζών. Τελευταίο σημείο που έχω να τονίσω είναι ότι η προτεραιότητα είναι η μείωση του κινδύνου. Αυτό ακούγεται καλά προφανώ, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και μια σημαντική υποσημείωση. Μέσω τη ρύθμιση μπορεί να ελέγξουμε τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε παντελώ τον κίνδυνο. Η ελπίδα, η πίστη σε αυτό, θεωρώ ότι οδήγησε σε ένα όλο και πιο περίπλοκο δίκτυο ε, κανόνων κεφαλαίου και σε, όποιο, σε όλο και πιο πολύ δυνατούς ε, μηχανισμούς ασφαλείας backstop που εφαρμόστηκαν στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο τα τελευταία χρόνια. Και όλα αυτά μπορεί να έχουν προκυκλικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις δημιουργώντας έναν ε, φαύλο κύκλο τέτοιων μηχανισμών. Συμπέρασμα. Η κρίση είναι ε, ένα χρονικό διάστημα για να λάβουμε άμεση δράση, αλλά όσο επίσης αποτελούν ευκαιρίες για πιο στρατηγική αναδιαμόρφωση. Και αυτή η κρίση δεν αποτελεί εξαίρεση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βράξουμε την ευκαιρία και να ξανασκεφτούμε το πώς προσεγγίζουμε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Και πιστεύω ότι μόνο αν το πετύχουμε αυτό, το τραπεζικό μας σύστημα θα είναι σε θέση να συμβάλλει στην απαραίτητη οικονομική ανάκαμψη, αντί να καταστεί τμήμα του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην κυρία Πέτιφορ. Αν Πέτιφορ. Mrs. Pettifor, could you please press the speak button? Thank you. Ah, sorry. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τους αξιότιμους ευρωβουλευτές που με συμπεριέλευαν στην συζήτηση αυτή. Θα τα πω ομά, μου επιτρέπετε. Έχουμε μάθει από την πρόσφατη κρίση του κορονοϊού ότι η έλλειψη προετοιμασία για κρίσεις που έχουν προβλέψει οι επιστήμονες μπορεί να μας σκοτώσει, όπως ε, για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή ή η κατάρρευση της βιοπικιλότητας. Μας έχουν προειδοποίησει ότι τέτοιες πανδημίες ήταν αναπόθευτες. Μας τα έχουν πει ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο καθηγητής Γκόλντιν και ο Μάικ Μάρχερσαν. Επίσης, στο βιβλίο μου, η περίπτωση της Νέας Πράσινης Συμφωνίας που δημοσιεύτηκε το 2019, το έλεγα ότι κινδυνεύουμε από τέτοιους κραδασμούς. Δεν ήξερα ότι θα είχαμε πανδημία, ήξερα όμως ότι είναι πολύ εύθραυστο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε στον ανθρωπισμό μας, την συμπόνια μας προς τα άλλα όντα, ε, ζώντα όντα να μας βοηθήσει. Μας είπαν ψέματα ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Μάθαμε επίσης από την κρίση του κορονοϊού ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να κινητοποιήσουν μέχρι 21 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα για να στηρίξουν τη... τα μη τραπεζικά ιδρύματα και το χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως Wall Street, το City και η Φραγκφούρτη. Μάθαμε επίσης ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να συγκεντρώσουν φόρους για να χρηματοδοτήσουν την σωτηρία των τραπεζών. Μάθαμε επίσης, όπως εξήγησε και η κυρία Καπορ, ότι τα ομόλογα αποτελούν τη σποδηλική στήλη του οικονομικού συστήματος και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν για να έχουμε ε, καλές εξασφαλίσεις. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του κορονοϊού είδαμε ότι ακριβώς ε, η απασχόληση είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει να συγκεντρωθούν ε, φόροι που με τη σειρά τους πληρώνουν τα ομόλογα τα οποία εκδίδονται για να δημιουργηθεί απασχόληση. Και ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι η δημιουργία απασχόλησης, είναι οι καλές θέσεις απασχόλησης και οι ισορροπημένοι προπολογισμοί. Τίποτα άλλο. Μάθαμε από τον ΩΣΑ ότι 7,6% είχαμε κατάρρευση του ΑΕΠ και ότι η ανεργία διπλασιάζεται, ότι στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ψηλή και ότι αναμένεται 20% στην Ελλάδα, 18% στην Ισπανία, 12% στην Ιταλία, 10% στην Γαλλία. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι άνεργοι λοιπόν. Τι δείχνει αυτό, αυτό που είπανε και άλλοι οικονομολόγοι σήμερα, ότι Υπάρχει η ικανότητα στην Ευρώπη και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ε, ικανότητα. Υπάρχει αδυναμία στην οικονομία τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την διεθνή και γι' αυτό τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά. Οι κυβερνήσει υποφελούνται από την πλήρη απασχόληση, γιατί όπω είπαμε, η πλήρη απασχόληση δημιουργεί φόρου. Αγοράζονται ομόλογα, τα οποία επενδύονται στην απασχόληση. Μάθαμε ότι ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε καλές θέσεις απασχόλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μαθήματα που έχουμε πάρει. Οι επιστήμονε γνωρίζουν ότι ο ανθρώπινο πολιτισμό κινδυνεύει να καταρρεύσει αν η θερμοκρασία του πλανήτη αυξηθεί πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Επίση, γνωρίζουν οι επιστήμονε ότι η θερμοκρασία μάλλον έχει ήδη υπερβεί αυτά τα νούμερα. Κι όμως εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε προ ακραίε καιρικές συνθήκες, κλιματική καταστροφή και αυτή η κρίση, η πανδημία θα είναι μια απλή γρατζουνιά. Οι οικονομολόγοι γνωρίζουν ότι κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση από διάλυση. Οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι μια προσπάθεια εδραίωση τη Ευρώπη. Οι πολιτικοί επίση γνωρίζουν ότι η αποτυχία τη Πράσινη Συμφωνία να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή έτσι όμως ώστε οικονομικά να μην ξεχνά και κανέναν, θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης. Όπως έγινε και με την κρίση του κορονοϊού, οι χώρες θα προσπαθήσουν μόνες τους να προστατεύσουν τον κόσμο τους. Γι' αυτό και αυτά που διακυδεύονται είναι πολύ μεγάλα. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η στόχη μείωση εκπομπών της Πράσινης Συμφωνίας με 55% μέχρι το 2030, που είναι τρεις φορές πιο γρήγορα από ότι την περίοδο 90 με 1990 με 2020 δεν φτάνει. Χρειάζεται πιο φιλόδοξη στόχη. Και οι επιστήμονες και οι πολιτικοί μάλλον γνωρίζουν ότι αν δεν εδρεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα κυριαρχεί στον κόσμο η ισχύ των ΗΠΑ. Και οι οικονομολόγοι ξέρουν ότι αν δεν υπάρξει η εδραίωση αυτή της Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος θα εξαρτάται από το αμερικανικό δολάριο. Το πρώτο βήμα λοιπόν που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έπανε και προηγούμενο μιλητή είναι να εκδώσει εξασφαλίσεις, δηλαδή ευρωπαϊκά ομόλογα τα οποία χρειάζονται και τα ζητούν οι κεφαλαίοι αγορές για να χρηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας και να σταματήσει πια εξάρτησή μας από το ρηκτά καύσιμα. Τέτοια ομόλογα μπορούν να συγκεντρώσουν ποσά όπως αυτά που συγκεντρώθηκαν για την κρίση του κορονοϊού. Το δεύτερο βήμα θα ήταν να σταματήσουν οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσωνα που είναι 250 δισεκατομμύρια το χρόνο και όπως έδειξε και ο καθηγητής Ερβά Στόρμο έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα των χωρών μελών περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο το τρίτο βήμα θα ήταν να εισάγουμε έναν φόρο για τον άνθρακα 75 ευρώ τόνο διοξιδίου του άνθρακα με αποτέλεσμα 270 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσια φορολογικά έσοδα κάποια από τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες των πιο φτωχών ε, νοικοκυριών που θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για την ενέργεια. Επίσης, η εταιρείε θα πρέπει να επωφεληθούν από την Πράσινη Σύμφωνία και το τέταρτο βήμα θα είναι αύξηση του εταιρικού φόρου. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι η έλλειψη προετοιμασίας για κρίσεις που έχουν προβλέψει επιστήμονες τελικά θα μας σκοτώσει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.